All right. Uh, uh, uh, Συνάδελφοι, όπως αναμενόταν κάποιοι φίλοι μας καθυστέρησαν, αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά να ξεκινήσουμε, διότι έχουμε δύο θέματα τα απόγευμα στο πρόγραμμά μας και θέλουμε να έχουμε κάποιο χρόνο, όχι απλώς για τις παρουσιάσεις, αλλά και για συζήτηση. Χαίρομαι που καλωσορίζω τα μέλη του πάνελ, τον κύριο Σμιτ από το Copenhagen Economics που θα μας παρουσιάσει τα απορίσματα της μελέτης αξιολογήσεις συνεπιών των αποτελεσμάτων μη δράσεως ή ελλειπού συντονισμένης άξος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της κρίσεως, καθηγητή Κόνορν Αλεξάνδρ από το Κέντρο για τη Χρηματιστική Ανάλυση και Πολιτική του Πανεπιστημίου του Cambridge, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη μελέτη διαχείρισης της κρίσης στο παρόν στάδιο. Την πρώτη εκδοχή την ετοίμασε πριν την κρίση και τώρα δοθήσεις της κρίσης είχε κάθε λόγο να ενημερώσει, να επικαιροποιήσει την έκθεσή του και προσβλέπουμε σε αυτή την παρουσίαση. Ο κύριος Σμίτ είναι πρώτος. Έχετε το λόγο. Thank you Um, I will uh, move straight into what I think is, um, a pretty um, challenging topic in this. Παρακαλώ, ακούτε καλά τα ελληνικά. Έχετε και να κάνετε ένα ανέβημα στην καμπίνα υπαριθμών 7 πίσω από το Προεδρείο, αν ακούτε καλά τα ελληνικά. Είμαστε στη διάθεσή σας. Ένα ανέβημα προς την καμπίνα υπαριθμών 7 πίσω από τον Πρόεδρο, αν μας ακούτε. Δεν είναι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 Στη μελέτη λάβαμε διάφορα στοιχεία υπόψη. Πρώτα την πρόληψη. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εμποδίσει τις ανισορροπίες που δημιούργησαν την κρίση. Μείωση και έλεγχο το δεύτερο. Τι έγινε να μειωθούν οι αρνητικέ συνέπειε τη κρίση. Από όταν ανέκυψε και τι κάναμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των χωρών που περνούν κρίση. Τι έκανε για πρόληψη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι πήγε στραβά. Στραβά πήγαν τα πράγματα, αλλιώς δεν είχαμε φτάσει εδώ. Τέσσερα στοιχεία. Έβλεπε που πήγαινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπήκε στην κρίση με ανοιχτά μάτια. Δεν άκουσε τις προειδοποίησεις διότι υπήρχαν τα προμηνύματα. Καταλαβαίνουμε τα βασικά αίτια της κρίσης. Και τα μέσα, αν τα δούμε από επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσης, ήταν αδύναμα και αυτά που υπήρχαν δεν χρησιμοποιήθηκαν. Οι συνέπειες δεν έχουν μοιραστεί όμορφα στις χώρες. αυτοί που λένε το μυστήριο της Ευρώπης, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ισπανία, Λοιπόν, και χειροτερεύει η κατάσταση. Και οι χώρες αυτές που είχαν πρόβλημα από όταν άρχισε η κρίση είχαν πολύ μικρή ανάπτυξη. Το ίδιο και στις βαλτικές χώρες. Για την υπόλοιπη Ευρωζώνη, Ηνωμένο Βασίλειο, μετά και Σουηδία, οι συνέπειες ήταν λιγότερο δραματικές. Υπάρχουν διαφορές στον φάση σοβαρότητα των προβλημάτων. Αυτό σχετίζεται με τις ανισορροπίες που δημιουργήθηκαν πριν από την κρίση. Όλες οι χώρες που έχουν προβλήματα σήμερα είχαν σημαντικέ αυξήσει όσον αφορά τις θέσεις των τρεχόντων εξόδων και τελικά δεν πήγαιναν και καλά ανταγωνιστικά. Όλα αυτά μπορούσαν να τα δουν πριν την κρίση. Ήταν ορατά σημάδια. Ήταν ορατά λοιπόν όλα. Γιατί δεν ακούστηκαν προειδοποίησεις. Υπήρχαν προειδοποίησεις. θα αναφέρω μερικά προμηνύματα. Από το 2001 και μετά βλέπαμε το αποθεματικά ότι τα στεγαστικά δάνεια ήταν στοιχείο κινδύνου και ο τραπεζικός τομέας έλεγε ότι οι προβλέψεις για ανάπτυξη ε, δεν σχετιζόταν με τον κίνδυνο, με τις ανισορροπίες. Ο ΣΑ προειδοποίησε τις απειλές που δημιουργήθηκαν στις αλίδες των στεγαστικών δανείων. Και τα δημοσιονομικά προβλήματα τα έβλεπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Εκοφήν. Όμως, παρόλα αυτά, υπήρχε εφησυχασμός με αισιοδοξία όπως η G7 των κεντρικών τραπεζών το 2007 που δήλωσαν και είπαν ότι η παγκόσμια οικονομία έχει τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη την τελευταία τριακονταετία και γίνεται ισορροπημένη. Και οι πρόσφατε εξελίξει στη χρηματοπιστωτική αγορά και το hedge fund συνέβαλαν σημαντικά στην αποδοτικότητα του χρηματοστικού συστήματο, δηλώσει ένα χρόνο πριν καταρρεύσει το σύστημα, όπως λέμε και. και οι προβλέψεις δεν ήταν σωστές των χρηματοστικών ιδρυμάτων. Επί σειρά ετών δούλεψα στον ΩΣΑ και ξέρω ότι συνήθως υπάρχει μια τάση για συνένεση. Οπότε εκείνοι που κάνουν τις προβλέψεις δύσκολο να προβλέψουν σωστά. Υπήρχε υποτίμηση στις τεχνικές εκθέσεις αφορά τον κίνδυνο. Και επίσημες εκθέσεις τα ανέφεραν εκλογηγός. Δεκαετία του 90 ακολουθήθηκε στη ΣΥΠΑ πολύ χαλαρή χρηματοστική πολιτική. και υπήρχαν αμφιβολίες όσον αφορά την, τον καθαρισμό των επιτοκίων. Και από το 2001 και μετά μέχρι την κρίση ήταν πολύ χαμηλά τα επιτόκια και τροφοδοτούσαν συνειδητοποιήσεις. τα ίδια σημάδια που έβλεπε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, αλλά με μεγαλύτερο, σε μεγαλύτερο ποσοστό. Ανισορροπία στη ΣΥΠΑ που ξεχύλισε και επηρέασε και την Ευρώπη και όσον αφορά την πραγματική οικονομία και το χρηματοστατικό τομέα. Και είχαν και βέβαια και συμφέρονται ευρωπαϊκές τράπεζες στην αγορά της Αμερικής. Οικονομική πολιτική, ελλείμματα στις περισσότερες χώρες, ακόμα και την περίοδο των παχιών αργελάδων. οι χώρες που αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα είχαν πολύ μεγαλύτερα ελλείμματα από τις υπόλοιπες. Και βασικά είχαν προβλήματα οι χώρες που είχαν μεγάλο πληθωρισμό. Κανονικά πρέπει να ακολουθήσουν πιο σφιχτή φορολογική οικονομική πολιτική για να δίνουν κίνητα στην οικονομία. Άρα οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν δεν ήταν καλές. Κυρίως στις χώρες αντιμετώπισαν προβλήματα. Δεν έδιναν τα αναγκαία κίνητρα και δεν ενίσχυαν επαρκώς την οικονομία. Είναι και θέμα ρύθμισης και εποπτεία. Ήταν ανεπαρκή. Κακή διαχείριση του κινδύνου. Οι εποπτικές αρχές αδράνησαν η ε, οι εκθέσει σε κίνδυνο των διατραπεζικών συναλλαγών ήταν μεγαλύτερη από ό,τι έπρεπε. Όσον αφορά τη ρύθμιση και τον έλεγχο, και εκεί είχαμε προβλήματα και κενά και αποτυχίες. Θα το συζητήσετε στην Επιτροπή. Να μπαίνουν πολλά χρηματοπιστωτικά μέσα στην ίδια κατηγορία κινδύνου και οι φορείς βαθμονόμησης φερεγγιότητας ίσως βαθμολόγησαν πολύ χαλαρά και κυρίως στον τομέα των στεγαστικών δανείων και των διαφόρων αξιογράφων. Δεν τα ταξινόμησαν σωστά σε με τον κίνδυνο. Ποιο ήταν το κόστος της μη πρόληψης. Τι εννοούμε με μη πρόληψη. Τι έγινε σε εθνικό επίπεδο, οικονομική πολιτική, σε εθνικό επίπεδο. και ρύθμιση χρηματοπιστωτικών αγορών, θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί δεν πήγαμε καλά. Το κόστος ήταν πολύ μεγάλο της ελληπούς πρόληψης. Ανεργία, απώλεια δεξιοτήτων των ανέργων, κεφάλαια που δεν χρησιμοποιούνται. Και Ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι μπορεί να χρειαστεί μια τραπεζική κρίση 5 με 7 χρόνια για να έχουν αποτελέσματα οι πολιτικές. Το ξέρουμε από τη Σκανδιναβία. Ξέρετε πόσο κοστίζει στην Ευρώπη αυτό. Κάναμε προβολές. Τις δημοσίευσε ο ΣΑΠ πέρσι. Ίσως χρειαστούμε 5 με 7 χρόνια από τώρα μέχρι ότου επιστρέψει σε κάποια αμαλή κατάσταση η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Απόλυα διψήφια όσον αφορά ποσοστό του ΑΕΠ θα είναι η απόλυση. Μείωση και έλεγχος μετά. Κάπως καλύτερα πήγαμε εδώ, όσον αφορά τη μείωση των αποτελεσμάτων. μακροοικονομική υποστήριξη ήταν καλή από τη στιγμή που αναγνωρίστηκε η κρίση. Μετά κυρίως το Συμβούλιο του Μαρτίου 2009 είχαν πολύ χαμηλά επιτόκια, τα πιο χαμηλά της δεκαετίας και κεντρικές τράπεζες υποστήριξαν τη ρευστότητα των εθνικών ιδρυμάτων μέσω αγοράς αξιογράφων και εμπόδισαν τιμή στον των να αυξάνονται στη φερικιότητα για τον έλεγχο της κρίσης, η Ευρώπη δεν είχε σύστημα να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις σε κρατικό επίπεδο. Είναι φανερά τα αποτελέσματα τώρα που μιλάμε. Είδαμε παρόμοιο φαινόμενο το 2007, τεράστια αύξηση ελλημάτων. Λόγω αυτομάτων σταθεροποιητών, χαμηλότερης φορολόγησης, μεγάλων δαπανών, κρατικών και αύξηση των δαπανών για την υποστήριξη της οικονομίας. Τα αποτελέσματα ήταν υπιότερα από ό,τι τον είπα, παρόλο που η κρίση ήταν ε, μικρότερη εμβέλειας από τον είπα. Και η χαλάρωση των φορολογικών πολιτικών και οικονομικών πολιτικών τώρα, εν συγκρίση με αρχές δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90, οι απώλειες ήταν μεγαλύτερες όμως εν συγκρίση με το μέγεθος της κρίσης, που και αυτή είναι μεγαλύτερη. Βάσει ιστορικών στοιχείων, Ίσως να είχε αυξηθεί η παραγωγή και η εκροή στην Ευρωζώνη αν είχαν χαλαρώσει κάπως τα φορολογικά μέτρα, κατά 1%. Ακόμα και τεράστια φορολογικά και οικονομικά κίνητρα δεν θα μπορούσαν να αποφύγουν την κρίση. Είχαμε τα χαμηλότερα ονομαστικά επιτόκια επί δεκαετής. Τα πραγματικά επιτόκια μειώθηκαν λιγότερο, γιατί μειώθηκε ο πληθωρισμός. Αλλά μειώθηκαν και τα επιτόκια αρκετά. Υπάρχει ένα επιχείρημα που το αναφέρω συχνά. Οι χώρες που έχουν πλεονάσματα τρεχόντος ισολογισμού ή καλύτερα δημοσιονομικά θα έπρεπε να δώσουν φορολογικά οικονομικά κίνητρα για να υποστηρίξουν την εσωτερική οικονομία. όπως η Γερμανία, Ολλανδία και άλλες χώρες. Προβάλλουμε τέσσερα επιχειρημάτα. Υπέρ και κατά. Η Γερμανία πρέπει να κάνει περισσότερα. Ήταν μεγάλο το πακέτο ενίσχυσης οικονομίας της Γερμανίας και κινήτρων. χρέος προς ΑΕΠ είναι πέρα από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και αν δούμε εκτιμήσεις του τι θα έκαναν περισσότερα κίνητρα στη Γερμανία, τι αποτελέσματα, η διαφορά είναι μέτρια. Έχουμε διαβάσει πολλές μελέτες. 1% του ΑΕΠ αύξησε τις η Γερμανία. Και συνέπειε σε Πορτογαλία και Ιταλία θα ήταν 0,1 του ΑΕΠ. Άρα υπάρχουν όρια όσον αφορά το πώς ε, μπορεί να βοηθήσει η Γερμανία τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Είναι πλούσια χώρα η Γερμανία, αλλά και γυράσκουσα. Θα έπρεπε να οικονομήσει κάποια χρήματα και να σε χώρε που μπορεί να χρησιμοποιήσουν καλύτερα, λένε. 2-3% θα ήταν το πλεόνασμα της Γερμανίας, προβλέπετε. Και ο μέσο 4 5% τελευταία 4-5 χρόνια. Αντεπιχείρημα που λέει ότι η Γερμανία προσέχει περισσότερο τα γερμανικά συμφέροντα. Η ΕΠΑ και η Ευρώπη, εταίροι της, Γερμανίας, θα πρέπει να εξάγουν περισσότερο, να εισάγουν περισσότερο, να εισάγουν περισσότερο, να εξάγουν λιγότερο. Άρα θα πρέπει η Γερμανία για να αντικαταστήσει τα χαμένα έσοδα να κάνει κάτι. Αυτό είναι θέμα ιδίου συμφέροντος παρά βοήθεια το πραγματικό κόστος όσον αφορά τη μείωση των συνέπειων είναι ότι δεν σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με προγράμματα σταθεροποίησης γιατί μη εκτός Ευρωζώνης το Διεθνές Μεσοδοτικό Ταμείο παρενέβη για να βοηθήσει κάποιες χώρες εκτός Ευρωζώνης. Όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα τώρα, έχουμε την Ελλάδα και κάποιες χώρες άλλες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουμε ρήτρα στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ρήτρα που απαγορεύει την παρέμβαση άλλων χωρών προς βοήθεια πασχούσης χώρας. Δεν υπάρχει σύστημα αυτόματης αλληλεγγύης και το σχήμα υποστηρίξεω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου συναρτάται με διάφορες δομικές αλλαγές και προσαρμογές του προπολογισμού της συγκεκριμένη χώρας. Και, και στη ΣΥΠΑ οι πολιτείες δεν μπορούν να δεχτούν βοήθεια από ομοσπονδιακό επίπεδο. Ούτε η πόλη από πολιτεία. Όλοι οι μηχανισμοί συναπαγόνται κόστος. Δημιουργείται πλαίσιο αντιμετώπιση κρίσεων τώρα. Αλλά υπάρχει ένα κόστος διότι δεν υπήρχε κάτι πριν από την κρίση. Ίσως αυτό να καθυστέρησε δράση σε κάποιες από χώρες που ανεμίχθησαν στην κρίση δεν ήξεραν τι να κάνουν. Να κάνουν κάτι, να μην κάνουν κάτι, να κάνουν πολλά. Δεν ήξεραν τι θα το θέλει. Όλα αυτά είναι εικασίε τώρα. Η έλλειψη δομή εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστέρησε η αδίποτε εφαρμογή αναδιάρθρωσης. Δεν είναι πρόβλημα όσον αφορά απώλεια εκροών από Ιανουάριο, Φεβρουάριο κλπ το κόστος είναι διαφορετικού είδους. Αυξημένα επιτόκια για κάποιες από τις εμπλεκόμενες χώρες, Υπάρχει πρόβλημα μεταδοσής των προβλημάτων. Αν δεν βρεθεί λύση για την Ελλάδα, θα γίνουν οι άλλες χώρες, Φερρυπίν. Τι μορφή θα έχει τελική λύση. οι πιστωτέ θα πληρώσουν το μαλλί ή κάποιο άλλος. Δύσκολο το περιβάλλον που δημιουργείται έτσι. Όλοι οι μηχανισμοί επιλύσεως των κρίσεων δημιουργούν κάποιο μπέρδεμα. Δεν έχω συγκεκριμένη πρόταση. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα αριθμό όσον αφορά το κόστος. Συμπέρασματά μου. Για να αποφευθεί το κόστος της ύφεσης είναι να μην μπει στην ύφεση. Ίσως είναι απρόσωπο σχόλιο, αλλά είναι αλήθεια. Όταν δημιουργηθούν και καταρρεύσουν τεράστιες ανισορροπίες, τι να κάνουν οι κυβερνήσεις. Όταν υπάρχουν τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα και αμφισβητούν οι χρηματοστατικές αγορές την αξιοπιστία μιας χώρας, ίσως κάποια μέτρα τόνωσης να είναι αντιπαραγωγικά. Άρα τα προληπτικά μέτρα υπήρξαν αδύναμα. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει μηχανισμό κυρώσεων που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Θα μπορούσαν όμως. Άλλαξαν μια φορά. Συζητείτε τώρα τι να κάνουμε γι' αυτό. Δεν αφορά εμένα αυτό. Εποπτεία και έλεγχος. Αυτό είναι εντολή των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων διότι υποβάλλουν οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων πλευρά τραπεζών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κάτι που επεξεργάζεστε. Εκ των υστέρων, έχεις μια εικόνα Μετά από όλα αυτά, η Ευρώπη έκανε αρκετά καλά, έλαβε καλά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε τα νομισματικά επιτόκια, αντέδρασε καλά και στήριξε τράπεζες αγοράζοντας αξιόγραφα υποστηρίζοντας τη θεραγκαιότητά τους. Με μονομένες κεντρικές τράπεζες θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό μεγαλύτερη δυσκολία και θα δημιουργούνται στρεβλώσεις αν η λύση έλαμβανε χώρα σε ε, κρατικό επίπεδο. Εδώ ωφέλησε η Ευρώπη, πρέπει να το τονίσουμε. Όσον αφορά τον έλεγχο και τη μείωση των συνεπειών, η αντιμετώπιση σε κρατικό επίπεδο είναι λάθος. Ευχαριστώ κύριε Σνέ Σμιτ. Και τώρα οι συνάδελφοι μπορούν να σχολιάσουν, να υποβάλουν ερωτήσεις. Περβάσου να ξεκινήσεις. Είναι η συγγήτρια. Merci, merci de cette présentation, euh, comme souvent venant de Copenhague. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση και χρήσιμη. Λέτε πολλά ε, στην ουσία ότι αν τα πράγματα πήγαν ε, καλά ε, ήταν επειδή δεν υπήρχαν εξωτερικές επιλογές ή επειδή υπήρξε ένα εξωτερικό σοκ. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν δύο τρόποι να προσεγγίσει κανεί το κόστο μη Ευρώπη. Η κατάσταση που ήταν πριν από το σοκ, δεδομένη τη ε, έλλειψη και έλλειψη δυνατότητα πρόληψη ή δυνατότητα παρέμβαση, όλα όσα θα μπορούσε να είχε κάνει και δεν έκανε. Και έπειτα υπάρχει ένα άλλο τρόπο προσέγγιση, που είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ε, το σοκ υπήρξε, κάναμε αρκετά πράγματα. Εσείς είπατε ότι η Ευρώπη αντέδρασε αρκετά καλά. Ε, τώρα, σε σχέση με την Ισπανία, λέγεται, αναφέρατε ότι ίσως όλοι δεν είχαν, αν είχαμε σεβαστεί το σύμφωνο στεθαρότητας, θα είχαμε μετριάσει επιπτώσεις αυτού του διτού σοκ, που ήταν ένα σοκ και της χρηματοπιστωτικής αγοράς και του εμπορίου. Δεν θα είχαμε 10% ανέργων, όπως διατρέχουμε τον κίνδυνο μέχρι στο τέλος του έτους. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα έκανε όλα καλά. Ανέβηκε στο πρώτο βήμα, στο πρώτο σκαλοπάτι του βήματος, στις 9 Αυγούστου και έλεγε ότι θα αντιμετωπίσει την κατάσταση. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2008 μείωσε τα επιτόκια, ε, τα επιτόκια και στη συνέχεια δεν μπόρεσε να περάσει το μήνυμα στις κυβερνήσεις ότι τα τοξικά προϊόντα δεν πρόκειται να εξαφανιστούν έτσι. Δεν ξέρω, δεν ε, προτίθεται να το κάνει, δεν ήθελε κλπ. Αλλά όσον αφορά την Επιτροπή, ειλικρινά δεν πιστεύετε ότι υπήρξε μια ιδιαίτερα βραδία αντίδραση και μια συνειδητοποίηση ότι χάσαμε έναν ολόκληρο χρόνο. Ο Πίτροπος τη Ιστορικής Αγοράς εξέδωσε ένα έγγραφο κατόπιν τίματος του Πρόεδρου Μπαρόζο, ο οποίος ε, ήταν στην ε, εκλογική εκστρατεία το Φεβρουάριο 2008 έλαβε λοιπόν την πρωτοβουλία να στάξει αυτό το έγγραφο. Αλλά μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008 για μένα ειλικρινά δεν συνέβησαν και πολλά πράγματα ή τουλάχιστον όχι αρκετά. Γιατί όσοι παρακολουθούσαν τα πράγματα από κοντά έβλεπαν ότι δεν πρόκειται απλώς για μια προσαρμογή της ε, αγοράς αλλά τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα από αυτό ή πιο σοβαρά και μετά από το Σεπτέμβριο του 2008 εκπονήθηκε το πρόγραμμα. Θεωρείτε ότι υπήρξε, ήταν η Ευρώπη αρκετά ενωμένη εκείνη τη στιγμή. Θεωρείτε ότι στον τρόπο που οι χώρες μέλη εκπώνησαν ε, σχέδια υποστήριξης, προγράμματα υποστήριξης των τραπεζών ε, χωρίς να καθορίσουν τους όρους, θεωρείτε ότι αυτό ήταν αρκετό. Γιατί είπαν, εντάξει, θα δούμε τι γίνεται όσον αφορά τον ανταγωνισμό εκ των υστέρων ίσως θα έπρεπε να είχαν υποθεί τα πράγματα εκ των προτέρων και οι μόνοι που θα μπορούσαν να το είχαν κάνει τότε ήταν οι Ευρωπαίοι. Γιατί αν ε, ο Σαρκοζή το έκανε για τις ε, γαλλικές τράπεζες, δεν ισχύει και για τους άλλους. Επίσης ε, αναφέρατε τους οίκους πιστοληπτικής ικανότητας. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση του ρόλου τους. Έγινε μια μεταρρύθμιση, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω, είναι αρκετό αυτό ή υπάρχει ένα θέμα εδώ ε, τελικά μήπως εκπροσωπούν ένα επιχειρηματικό μοντέλο στον τρόπο που λειτουργούν ε, ε κατασκευάζοντας ορισμένα προϊόντα τα οποία πούλησαν στη συνέχεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές ε, χωρίς αυτά τα προϊόντα να είναι απολύτως ασφαλή. Και βεβαίως τον ε, αμφίβολο ρόλο που διαδραμάτισαν στην ελληνική κρίση. Πώς το εκτιμάτε? Θα προσπαθήσω να απαντήσω. I um, uh, Αφορά τα εξωτερικά σοκ. Ε, ε η κρίση αναδύθηκε τον ε, Οκτώβριο 2008 συντυπία κατάρρευσης μεγάλης επενδυτικής τράπεζας με, με σημαντικές διασυνδέσεις με, μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματο, με μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Νομίζω οι υποκείμενες αιτίες Ή για να το πω διαφορετικά, ο λόγος που πυροδότησε αυτή την κρίση ήταν οποιαδήποτε άλλη κρίση που, ή, οποιαδήποτε άλλη κρίση ξεκινάει με μία χρηματοπιστωτική κρίση. Γιατί οι επενδύσεις ε, τελικά συνδέονται με αυτές τις ε, φούσκες των χρηματοπιστωτικών της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Ο λόγος που πυροδότησε τελικά το 2008 ήταν αυτό το εξωτερικό σοκ που τελικά μεταδόθηκε στην ε, Ευρώπη. Και κατά κάποιο τρόπο οι ανισορροπίες που δημιουργήθηκαν σε ορισμένες από αυτές τις χώρες θα είχαν εκφραστεί εν πάση περιπτώσει. Έτσι λοιπόν δυσκολεύομαι να δω οποιαδήποτε χώρα, γιατί απλούστατα η κρίση αυτή στην Ευρώπη δείχνει ότι οι χώρες αυτές ήταν εκτεθειμένες στο σοκ αυτό. Η δική μου εντύπωση είναι ότι οι ισπανικές τράπεζες δεν θίγησαν από την κρίση στις πολιτείες σε αντίθεση με τις γαλλικές ή τις γερμανικές τράπεζες και τράπεζες του, της Μεγάλης Βρετανίας θίγησαν, αλλά όχι οι ισπανικές ε, τράπεζες. Πράγμα που δείχνει σε μένα ότι οι λόγοι στην Ισπανία, στην Ελλάδα ή την Πορτογαλία συνδέονται με κάτι που συμβαίνει στις ίδιες τις χώρες. Δεν ξέρω αν αυτή είναι μια ικανοποιητική απάντηση. Τώρα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νομίζω ότι προσπάθησα να πω ότι όλοι ότι ήταν πολύ πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο ε, εγώ στην νότητά μου ήμουν στον ΟΣΑ σε μια επιτροπή όπου κάποια προεξάρχουσα προσωπικότητα ρώτησε κάποιον άλλον από τη ΦΕΔ πότε θα αυξήσετε τα επιτόκια από το 1 στο 5% γιατί έχετε, αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα και χρειάστηκε να περάσει πολλής χρόνος για να γίνει αυτή η αύξηση επιτοκίων. Ε, νομίζω το έκανε λίγο πριν την κρίση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, να, δεν ήταν σε ε, καλή θέση με τα χαμηλά επιτόκια. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά τα όργανα βλέπουν από τη μία να αναδύεται το κίνδυνο του πληθωρισμού και θεωρούν ότι ίσως δεν έχουν απόλυτη συνείδηση των κινδύνων που φέρουν οι οικονομικέ ανισορροπίες. Πολλές φορές λοιπόν υπάρχει μια δυναμία αναγνώρισης αυτού του κινδύνου, δυναμία αξιολόγηση του μεγέθους του κινδύνου. Ίσως δεν ήταν ε, η σωστή αντίδραση στην εποχή εκείνη δεδομένων των ανισορροπιών. Μπορεί να το ισχυριστεί κανείς. Ε, αν θέλει κανεί να κρατήσει χαμηλά τα επιτόκια και να είναι κάτι για τη μόχλευση, νομίζω ότι το, ο προγραμματισμός ήταν ίσως εσφαλμένος οι μεγάλοι επίσημοι οργανισμοί και η Επιτροπή ε, άργησαν στη διαπίστωση, στη διάγνωση της κρίσης και επίσης δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν έγκαιρα. Ο ΩΣΑ άργησε το 2008. Μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο στη διάγνωση της κρίσης. Ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2009 εγώ θα έλεγα δεδομένη της έλλειψης αυτής της ε, διάγνωσης συνειδητοποίησης, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι ταχύτερη η απόκριση. Αλλά συμφωνώ μαζί σας όσον αφορά το εξής. Και ε, αναφέρομαστε σχετικά στην έκθεση, δεν μπόρεσα να σου παρουσιάσω σήμερα, αλλά αν ε, ξεκινήσουμε τις δύο σημαντικές δράσεις που αναλύθησαν στο εθνικό επίπεδο επιπρόθεστα προς τα ε, οικονομικά ερεθίσματα, η ενίσχυση ε, έθεσαν ορισμένες προκλήσεις προς την χώρια αγορά Διάβασα κάποιες έρευνες όπου αναφέρουν ότι τα πακέτα των τραπεζών ήταν, είχαν έλλειψη συντονισμού, είχαν πολλά χάσματα, αλλά και ένας από τους λόγους που δεν ήταν πολύ ουσιαστικά ήταν το γεγονός ότι οι αυξήσει στα ασφαλιστικά συστήματα θα ήταν πιο προβληματικά αν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες είχαν αποφασίσει να κάνουν αυξήσεις στα ασφαλιστικά συστήματα χωρίς περιορισμούς. Το γεγονός ότι κάποιες αλλαγές Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε αυτό. Τελικό αποτέλεσμα. Οι περισσότερες τράπεζες δημιούργησαν την εντύπωση ότι παρέχουν πολύ μεγάλη κάλυψη στους καταθέτες. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να κινητοποιηθεί, να θέσει προσανατολισμού. Δεν έκανε κάτι τέτοιο και αυτό ήταν λάθο. Το ίδιο και με την αυτοκινητοβιομηχανία. Στη μελέτη θέλαμε να δούμε αν υπήρχε μεγάλο κόστο ε, στην πραγματική οικονομία, μεγάλες τρευλώσει στην εσωτερική αγορά. Προφανώ όταν κάποιε κυβερνήσει προσπαθούν να κάνουν αναδιάθρωση σημαντικών αυτοκινητοβιομηχανιών, θέτοντας όρους, δηλαδή λέγοντα, αν θέλετε αυτό το παραδάκι, και κρατικέ εγγυησει πρέπει να ευνοείται θέση απασχόληση στη χώρα μας. Δεν έπρεπε να γίνεται αυτό όμως. Όμως, να πούμε ότι αυτό δημιουργεί μεγάλο κόστος για την Ευρώπη, αμφιβάλλω. Δεν νομίζω ότι ήταν ωραίο και καθαρό. Παρ' όλα αυτά όμως δεν δημιούργησε σημαντικές ε, δαπάνες. αν καθυστέρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι, διότι ε, παρεξήγησε τη συγκυρία, την υποτίμησε, ασυντόνιστες οι δράσεις για υποστήριξη τραπεζών κλπ. Τι λέμε στο κείμενο. Βλέποντας το πώς έχουν εφαρμοστεί διάφορες οικονομικές πολιτικές στην Ευρώπη. Πόσο γρήγορα θα κινούνταν οι χώρες αν έπρεπε να αποφασίσουν εκ των προτέρων επί των συνθήκων. Δηλαδή, ε, έχεις από τη μια πλευρά ταχύτητα, από την άλλη ουδετερότητα, αν θέλετε. Οι χώρες εφάρμοσαν μέτρα για να αυξήσουν την εσωτερική ζήτηση των οικονομιών τους. Ένα καλύτερο πακέτο θα προσπαθούσε να αυξήσει τη ζήτηση πιο ουδέτερα και για όλη την Ευρώπη. Αυτό θα χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο. Τελευταίο ερώτημα, για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Uh, για τους ε, οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ε, ικανότητας είχα θέσει το ερώτημα. Δεν είδα τη δουλειά σας, για να είμαι ειλικρινής. Επί χρόνια και χρόνια, καιρούς και ζαμάνια συζητάμε αυτό το θέμα. Ποιον εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις αυτοί φορείς που εκδίδουν ε, αξιόγραφα έτσι επενδυτές. Το ίδιο ισχύει και για τους λογιστές και για κάποιες επενδυτικές τράπεζες. Το ποιος εξυπηρετεί ποιον πρέπει να ε, εξεταστεί. Αυτό είναι ένα θέμα. Όλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. ε, ομαδοποιείτε τις χώρες σε 7 ομάδες από ό,τι βλέπω εδώ. Βλέπετε εφικτό τρεις ομάδες από ε, τον βόρειο αρκτικό κύκλο να τις βάλετε σε μια χωριστή ομάδα. Δανία, Σουηδία, Φιλανδία. Με παράλληλες εξελίξεις. Λίγο πολύ. Η Δανία είχε ένα πρόβλημα στη δεκαετία του 80, την, την τιμή της πατάτας και το ίδιο είχαμε και εμείς στη δεκαετία του 90. Άρα, νομίζω ότι οι επιπτώσεις ήταν τόσο σοβαρές τελικά και νομίζω ότι όλες οι εταιρείες αυτών των κρατών έχουν καλή πρόοδο. Άρα θα έχουμε μεγάλους σταθεροποιητές νομίζω αυτόματος. Οι οικονομίες ε, δεν υπέσταν τόσο μεγάλα πλήγματα. Υπήρχαν, όπως είπα, εξαιρέξεις. Και εμένα μου τελείωσε το μαγικό φίλτρο. Το μαγικό φίλτρο. Ίσως πρέπει αυτές και τις χώρες λοιπόν να συμμεχωριστούν. Για, τις, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Πριν από 6-7 χρόνια έχει εκφραστεί μία πρόταση να αυτορυθμίζονται. Η Caesars το είχε πει αυτό τότε. Σήμερα η Standard Poor's υποβάθμισε την Ισπανία και όλος ο κόσμος αντέδρασε. Μα αν είναι τόσο απρόβλεπτα τα πάντα και δεν τους πιστεύει κανείς, γιατί τους, τους πιστεύει η αγορά, γιατί να προκαλούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Θα ήταν καλό νομίζω να δούμε και αυτό το ζήτημα. Και τώρα πια έχει λήξει η κρίση. Τέλειωσε. Πρόεδρος, εγώ θα καλέσω και τους συναδέλφους από τη Φιλανδία να μιλήσουν στην υπόθεση αυτή. Ναι, ευχαριστώ και εγώ, όπως ούλε είχα μια αντίστοιχη ερώτηση, αλλά από μια διαφορετική έποψη. Μιλάτε για κάτι κατηγορίες όπου η Σουηδία και το ρεμένο Βασίλειο έχουν σταθεί στα πόδια τους ακόμα, δεν έχουν καταποντιστεί, αλλά βρίσκονται και έξω από τη ζώνη του ευρώ. Μήπως είναι αυτός ο λόγος τελικά. Και επίσης θα μπορούσατε να κοιτάξετε λίγο περισσότερο ποια θα μπορούσε να είναι η μετέπειτα κρίση. Και τι είδου ε, φούσκες μπορούμε να περιμένουμε για το μέλλον. Απάντηση. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ νόημα να κάνουμε τι συγκρίσει κατά αυτόν τον τρόπο, να βάλουμε την Δανία δηλαδή με τι άλλε χώρε. Γιατί είναι de facto μέλο τη Ευρώπη, ε, δεν έχουμε κειμενόμενη ισοτιμία, έχουμε μια σταθερή νομισματική πολιτική. Και ενώ άλλες χώρες έχουν ε, υποβαθμίσει τα νομίσματά τους, το τελευταίο διάστημα προς το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπορεί να μπει στην ίδια ομάδα η Δανία. Ταυτόχρονα οι ίδιες χώρες έχουν σημαντική αύξηση στο στο τελευταίο διάστημα. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει μια ιστορία που χαρακτηρίζει, θα έλεγα, ιδιαίτερα τα κράτη του Βόρειου Αρκτικού Κύκλου εδώ πέρα. για τις υπηρεσίες, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Και αυτοί, όπως και άλλοι επενδυτές, έχουν σαν χαρακτηριστικό να εντοπίζουν κινδύνους και να ε, δραστηριοποιούνται όταν ε, μάλλον θα έπρεπε να γίνεται το ανάποδο. Ε, εν πάση περιπτώσει όμω θα πρέπει να δούμε αν αυτοί οι οίκοι αξιολόγηση ψηφιακή ικανότητα συνεργάζονται με ε, τι κυβερνήσει των κρατών μελών και με τα, τις κεντρικές τους τράπεζες. Πολλές φορές έχω συζητήσει από τον ε, οίκο αυτών με εκπροσώπους που με ρωτούσαν κάθε χρόνο πώς πάει η Δανία, πώς πάει η οικονομία της Δανίας κλπ. Εντάξει, μετά τα σάφισα στην πείρα μας. Σταμάτησα. Ο τελικός λοιπόν επενδυτής μπορεί να ενημερώνεται ότι θα πρέπει να επενδύει με ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Και όσο υψηλότερη είναι η επιστοληπτική αξιολόγηση, τόσο χαμηλότερο θα είναι το ποσοστό το οποίο θα αναμένει. Απλώς υποκαθίσταται η αξιολόγηση του ιδίου του επενδυτή. Άρα μήπως είναι απλώς μια ανάθεση σε εξωτερικό παράγοντα της αξιολόγησης του κινδύνου και τίποτε περισσότερο. Ναι. και μήπως δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων εφόσον υπάρχει αυτή η συνεργασία με τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις. Δεν έχουν τον ίδιο ρόλο εναντί των κρατικών χρεών αφενός και των χρεών του ιδιωτικού τομέα αφετέρου αυτή η οίκη αξιολόγηση πιστολογικής ικανότητας. Αυτό πρέπει να το διαφοροποιήσουμε. Because they are not involved in the actual issuance of paper. Όχι, όχι, απλώς δεν έχουν, ε, δεν έχουν αυτή τη λειτουργία, αυτό είναι όλο. Οι ερωτήσεις δυστυχώς είναι εκτός μικροφώνου. Μα του, η Σίζαρ το εξέτασαν όμως. Και θεώρησαν ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω ρύθμιση. Το σημειώνω, λέει ο κύριος Νέα Σμιτ. Θα το περιλάβω στην έκθεση εφόσον χρειάζεται. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μάλλον προς την αντίστροφη κατεύθυνση η αξιολόγηση. Τι ερώτηση είχατε εσείς? Ναι, αλλά κοιτάξτε να σας πω, εάν λέτε ότι η Βρετανία και η Δανία και η Σουηδία είναι στο καλύτερο επίπεδο ενώ βρίσκονται έξω από τη ζώνη του ευρώ, μάλλον δυσίωνες προβλέψεις μας κάνετε, δηλαδή τι να φανταστούμε ότι μας περιμένει. Και ποιοι θα είναι οι επόμενοι λόγοι για την προσεχή κρίση. Λοιπόν, δημοσιεύθηκε κάτι πριν από κάποια κρίση, δημοσιεύθηκε κάποιους μήνες πριν μια έκθεση και διάβασα ένα ωραίο βιβλίο από τον Σύρο, έναν Αμερικανό. Ανάλυσε όλες τις σχηματοστατικές κρίσεις από το δεκαετία, από το 1880. Αξίζει να το διαβάσετε το βιβλίο. Διότι όλες οι καταστροφές της χρηματοδοτικής αγοράς έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό. Ο κόσμος είναι... εφευρέθηκαν τεχνικές, εμφανίστηκαν ε, νέοι κίνδυνοι κλπ. Τέλος 18 αιώνα, 19ου αιώνα, τα χρήματα πήγαν στον ηλεκτρισμό. Όλες οι ηλεκτρικές εταιρείες χρεοκοπούσαν. Οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι βιομηχανίες είχαν κέρδη. Δεκαετία του 20 η παγκόσμια η οικονομία έβγαλε τον ίδιο όρο, νέα οικονομία, όλο την ίδια λέξη χρησιμοποιούσαν, νέα οικονομία κάθε φορά. Για 15-20 χρόνια δεν συμβεί ξανά αυτό, διότι αυτοί πρέπει να τι αποφάσει θυμούνται ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Και μετά από 25 χρόνια το ξεχνούν αυτοί πλέον τι αποφάσει και επαναλαμβάνει το κύκλο των λαθών. Πολλά μπορούν να γίνουν όμω. Και εμεί έχουμε προτείνει στην εκθεσούλα μα κανόνε που μπορούν να βελτιωθούν όπως έγινε κατά το παρελθόν. Και μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε για να εμποδίσετε κι άλλη καταστροφή. Να επανελθεί στο μέλλον μια καταστροφή. Η ΚΕΙ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ερώτημά μου έχει δύο μέρη. Πρώτον, πώς ξέρουμε ότι συγκρίνουμε μήλα και μήλα αντί μήλα μαχλάδια. Πολλοί καθορίζουν διαφορετικά την ανεργία. Στην ΟΒ αλλάξαμε τον ορισμό, ανάλογα με το τι θέλουμε να δείξουμε. Ανησυχώ λοιπόν, όταν βλέπουμε συλλογικά τσιματοποιημένα στοιχεία για να δούμε ποιος θα πάει καλά και ποιος άσχημα, καλύπτεται μια τεράστια εικόνα που είναι πίσω από τους αριθμούς. Αν δεν καθορίσουμε τι αριθμούς ψάχνουμε, τότε να κάνουμε συγκριτική ανάλυση μας δίνει ασφαλμένη ανάλυση. Υπάρχει μηχανισμός για να έχουμε τυποποιημένα στοιχεία, μήτρες στοιχείων κλπ. Θέλετε ή σαν οικονομολόγος χαιρόσαστε ότι βρείτε μπροστά σας να πάρετε που σας δίνουν τα κάτι μελη Η Eurostat προσπαθεί από πλευρά δημοσίου χρέου να ξανακαθοριστούν τα στοιχεία τα αριθμητικά. Ξέρω στη δική μου περίπτωση έχουμε τεράστια, τεράστιο έλλειμμα του ισολογισμού και τα στοιχεία δεν είναι καλά γιατί δεν βγαίνει άκρη όταν κάνουμε την, ε, τους υπολογισμούς. Έχετε μια διαφάνεια. Λέτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σχεδιαχεί για προγράμματα ω τύπου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ερώτηση. Θα έπρεπε να έχει σχεδιαστεί έτσι. Απάντηση. Ανεργία. Τα, ποσοστά ανεργίας που χρησιμοποιούμε στη μελέτη είναι τα τυποποιημένα ποσοστά. Αυτά που χρησιμοποιεί ο ΣΑ. Όταν βλέπετε τις επίσημες προβλέψεις είναι επίσημα ποσοστά ανεργίας των κρατών μελών, που καμιά φορά σε επίπεδο κρατών μελών όπω είναι το Ηνωμένο Βασίλειο αλλάζουν για κάποιου σκοπού τα στοιχεία. Και μετά έχετε τυποποιημένα στοιχεία διεθνή που είναι πια αντικειμενικά για το χρέος. Έχουμε ανάληψη υποχρεώσεων εκτός ολογισμού που δεν μπορούμε να το... είναι διαφορετικό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα, όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία, χρειάζεται έρευνα και αυτό. Στη μελέτη μας έπρεπε να αρκεστούμε με τα επίσημα στοιχεία που μας διέθεσαν. βλέποντας ιστορικές αξιολογήσεις υπολογισμούς. Υποστήριξη για το τραπεζικό τομέα. Εκ των υστέρων, ε, το τελικό κόστος ήταν χαμηλότερο από τους υπολογισμούς. Με προβλέψεις στη Σουηδική κρίση τελικά μετά τα μέτρα βγήκαν κερδισμένες οι τράπεζες. Και στη ΣΥΠΑ ήταν θετικά τα αποτελέσματα. Ίσως τα αριθμητικά στοιχεία να είναι υπερβολικά, να είναι πιο μεγάλα από ό,τι έπρεπε. Το χρέος όμως συμπεριλαμβάνει χρηματοδοτικές επενδύσεις στοιχεία ενεργητικού, κάτι που αφορά τις τράπεζες που ελπίζουμε τελικά αυτά τα αξιόγραφα στο μέλλον να αυξήσουν την αξία τους. Άλλωστε, Περβόν, Ναι, ήθελα να πω κάτι, μια διευκρίνηση όσον αφορά τις εργασίες. Μια διευκρίνηση για τι εργασίε του ΣΕΖΑΡ. Αυτό στο οποίο αναφέρει το Όλι Σμιτ είναι τη ε, Γιούσκο οι εργασίες που μιλούσε για ένα κώδικα ε, καλή συμπεριφορά που θα σπίσει το 2004 και που στη συνέχεια επικυρώθηκε από τη Σέζαρ. Εν πάση περιπτώσει, το σημείο αυτό εκκίνηση είναι η καταγραφή από τη Σίζαρ ενό κώδικα συμπεριφορά που είχε η Γιούσκο συστήσει, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Πρόεδρο, θα τα δούμε αυτό στο τέλος σα. Και εκεί που λέγαμε ότι βγήκαμε από την ε, τραπεζική κρίση, φαίνεται να πέφτουμε σε, ένα, σε μια κρίση εθνικού χρέου. και θα ήθελα εσεί να μα εξηγήσετε, να μα πείτε πώ κρίνετε την κατάσταση και πώς ίσως να έχει και μεταδοτικότητα σε άλλα κράτη. Πρώτον ερώτημα. Σε μερικά χρόνια δηλαδή τι μπορούμε να περιμένουμε. Και δεύτερον, σε σχέση με το εθνικό χρέος πάλι. Πρέπει πράγματι να χρησιμοποιούνται οι εκτιμήσεις των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Δεν υπάρχουν οργανισμοί εδώ επίσημοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν υπάρχουν δεν κάνουν τη δουλειά του. Που θα είναι και πιο ουδέτεροι ίσως και πάντως δεν θα έχουν τον πειρασμό της κερδοσκοπία. Το ζώο... Και δεν ε, υπάρχει δυνατότητα διακυβέρνησης ε, έτσι ώστε να καθοδηγήσει μια χώρα πέρα από την, έξω από την κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση. κάποιο συντονισμό, κάτι τέτοιο, εν περιπτώσει. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Αν ερχόταν ο Μπαρόσο να σας πει τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στην Ευρωζώνη, για το Ευρώ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Τι είδους δημοσιονομικές και οικονομικές βιοπολιτικές μπορούμε να αναπτύξουμε από κοινού. Για την κρίση του εθνικού χρέους. Ναι, δεν είναι σαφές αν ε, φταίνε οι ίδιοι. Και ναι, εάν υπάρχει συνεχιστή κερδοσκοπία θα πάνε όλα στραβά. Έχω ένα φίλο που διαχειρίζεται ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο δανέζικο και είπε ότι θα, το καλύτερο που θα μπορούσαν να κάνουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία θα ήταν να μείνουν μέσα στο ευρώ και να επιμείνουν για το ευρώ και να, να είναι ο πυρήνα του ευρώ και όχι να αποχωρήσουν, γιατί αν αποχωρήσουν πάλι θα μείνει το χρέο του σε ευρώ. Δηλαδή, ακόμη μεγαλύτερε δυσκολίε θα έχουν να ξεπληρώσουν το χρέο. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή, ό,τι και να πούμε. Ό,τι μηχανισμός και να αναπτύσσετε τώρα, από την Επιτροπή, κάτι μέλη, το Διεθνές Μοσπονδικό Ταμείο, την Κεντρική Τράπεζα, να είμαστε, ανά πάσα στιγμή, να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη τα οποία φταίνε για τα σοβαρά προβλήματα θα υποστούν τις συνέπειες και ταυτόχρονα θα έχουν και αρκετή υποστήριξη για τον πρώτο τουλάχιστον χρόνο, που μάλλον θα αρκεί, και θα υποστηριωθούν να καταβάλουν επιτόκια, ναι, μένα, ε, κυρωτικά, αλλά πάντως όχι ασήκωτα. Και όταν μιλούμε για εθνικό χρέος, Γιατί πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων και του εθνικού χρέους. Είναι τελείως διαφορετική κατάσταση, όροι κτλ. Μία χώρα, μόνο εάν δεν θέλει να πληρώσει, μπορεί να κριθεί αφαιρεγγύο. Όχι αν δεν μπορεί, γιατί η Ελλάδα τώρα δεν μπορεί. Το θέμα είναι μόνο αν δεν θελήσει να πληρώσει. Μπορεί μια χώρα να κριθεί ως αφαιρέγγια. Η βούληση δηλαδή είναι το κριτήριο σε περίπτωση εθνικού χρέους. Και αυτό ένας πιστολεπτική, αξιολόγηση τη πιστολεπτική ικανότητα δεν μπορεί να το δει αυτό, ούτε τον ενδιαφέρει. Κάνει διαφορετική υπόθεση. Άλλο μια επιχείρηση, άλλου τύπου ε, χαρτοφυλάκιο έχει ενεργητικό, παθητικό, έσοδα, έξοδα. Επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο ενδεχομένως κρίνεται ανεπαρκές. Και τότε μπορεί στην επιχείρηση, στον επιχειρηματία να πει πλήρωνε κι άλλα, αλλιώ πα φυλακή. Στο κράτο όμω δεν μπορεί να το αυτό, στο εθνικό χρέο. Άρα, πέραν των οίκων πιστολεπτικής, αξιολόγησης πιστολεπτικής ικανότητας, πρέπει ο κάθε κράτος ή κάθε διεθνής οργανισμός να έχει τη δική του αξιολόγηση. Το μόνο που μπορεί να κάνει ένας τέτοιος οίκος αξιολόγησης πιστολεπτικής ικανότητας είναι να συστήσει στους μεγάλους επενδυτές με τη βαθμολόγηση από το ΑΑ στο Β κτλ. τις τιμές που μπορούν να χορηγηθούν για το δανεισμό. Ο ρόλος όμω είναι διαφορετικός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι οίκοι αξιολόγηση πιστολοπτική ικανότητας έχουν ιδιαίτερο ρόλο στην αξιολόγηση μιας επιχείρησης, αλλά καθόλου τον ίδιο ως προς το εθνικό χρέος μιας χώρας. Και αν εμφανιζόταν ο Μπαρόσο που λέτε πριν, Εάν η Επιτροπή, παραδείγματι, καταθέτει τάσεις και για αξιολόγηση από τους ομολόγους ε, και για ε, εκ των προτέρων ε, κρίση των προτάσεων ή των μέτρων, φιλόδοξο μου φαίνεται, υπερβολικά ίσως φιλόδοξο, ίσως μη ρεαλιστικό, το ΕΚΟΦΗΝ, το Συμβούλιο, μάλλον θα βρεθούν αναγκασμένα να να ξεπροστιάζουν δημόσια όποιο κράτος βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Εκεί θα καταλήξουμε τελικά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της απόψινής συνεδρίασης. Ο κύριος Αλεξάνδερ από το Cambridge, καθηγητής, για να μας μιλήσει για τη διαχείριση της κρίσης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και τους οργανωτές εδώ που με καλέσαν και πάλι να παρακολουθήσω την συνέχεια μιας μελέτης που είχαμε ξεκινήσει το 2007 το φθινόπωρο. Μόλις είχε αρχίσει να σκάει μύτη η κρίση. Όταν ε, η κρίση στα subprime, στα δάνεια, είχε αρχίσει να επεκτείνεται στις Ηνωμένε Πολιτείες και ε, έχαναν τις εγγυήσεις τους, τις εμπράγματες, οι τράπεζες ε, το φθινόπωρο, όπως είπα, το 2007. Ξεκινήσαμε μια μελέτη των ε, λόγων που οδήγησαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε αυτό το πρόβλημα. Και εδώ στην παρουσίασή μου αυτό που θα ήθελα θα ήθελα να σας εξηγήσω και βέβαια τη συνέχεια της μελέτης μας, τη μελέτη για τη διαχείριση, αλλά και το τι άλλο θα μπορούσε να γίνει από εδώ και μπρος. Συστάσεις δηλαδή. Κοιτάμε λοιπόν τις επιπτώσεις της κρίσης, ε, τι ε, τις ρίζες του κακού και διαπιστώνουμε ότι δεν προσφέρουν τα μοντέλα διαχείρισης κινδύνου επαρκείς ε, δικλίδες ε, για την αποφυγή των κινδύνων για τις τράπεζες. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ρευστές κεφαλαιοχικές αγορές και υπερσυνοριακές ροές κεφαλαίων να μην μπορούν να εμποδίσουν το αυτόματο πάγωμα κεφαλαίων και αγορών, όπως έγινε, όπως είπα, σχεδόν αυτόματα μέσα σε μια νύχτα το 2007 το φθινόπωρο. Επίσης θα πρέπει ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα να δείχνουμε σε κανονιστικά μοντέλα που στηρίζονται στις αγορές, ε, έλεγχο συστημικών κινδύνων από τα αριθμιστικά πρότυπα διότι αυτά τα αριθμιστικά πρότυπα που ε, είχαν εφαρμοστεί 7-8 χρόνια πριν από την ε, εμφάνιση της κρίσης ήταν ευαίσθητα, ε, τίναν νους στις ανάγκες της αγοράς, δηλαδή ήταν κυρίως στηριγμένα στην αγορά. Και παράδειγμα είναι η Βασιλεία 2, παρότι δεν προκάλεσε κρίση, το πρότυπο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η συμφωνία αυτή ήταν μέρος του προβλήματος και στη βάση των, των χρηματοπιστωτικών αγορών. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο προσαρμόζεται η ρύθμιση από τα ρυθμιστικά όργανα, τις ρυθμιστικές αρχές, μετά, στη φάση της καινοτομίας, μετά την κρίση δηλαδή, που μπορεί ενδεχομένως και να εντείνει τις εξωτερικεύσεις, εξωτερικότητες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει οι, ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις να είναι πάντοτε στην επικαιρότητα και να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες, γιατί βέβαια το να παραμείνουμε στάσιμοι σημαίνει και βέβαια ωφέλη, αλλά και μεγάλους κινδύνους όπως έγινε με τα δάνεια. Είδαμε ότι και η Επιτροπή της Βασιλείας αλλά και άλλοι διεθνείς οργανισμοί απέτυχαν στον εντοπισμό των κινδύνων σε μια αρχική φάση και σε μια έγκαιρη φάση καλύτερα και ότι υπήρξαν κάποιες εκθέσεις από ορισμένου που κατά ύποπτο τρόπο επεσήμεναν ότι υπάρχει αύξηση στις τιμές ε, των ακινήτων, ενώ φαίνεται ότι δεν εκρίθη αρκετά σοβαρό αυτός ε, πρόβλημα από τις ρυθμιστικές αρχές. Και γιατί η εντολή τους για την νομισματική πολιτική περιοριζόταν μόνο στην, στον πληθωρισμό, στις τιμές λιανικής και δεν μπορούσαν να λάβουν υπόψη ευρύτερη εικόνα των τιμών, φερρυπίν τιμές των ακινήτων το σώμα Λαμφαλούση, η Επιτροπή Λαμφαλούση, που είχε έναν στόχο αντίστοιχο όταν συναισθήθη, πάλι δεν μπόρεσε να αξιολογήσει τον κίνδυνο ε, που απειλούσε το ευρωπαϊκό σύστημα και ιδιαίτερα η Επιτροπή επίπεδου 3, διότι παρακολουθούσε ρυθμιστικό πρότυπο στηριζόμενο στην αγορά, ακατάλληλο για την ανάληψη μέτρων ε, σε περίπτωση περιορισμού των δυνατοτήτων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και βεβαινή ανταγωνιστικότητα με τι ΗΠΑ. Οι δε εθνικέ αρχέ εποπτεία δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στι ανησυχίε και τι ανάγκε για ε, ορθολογική συμπεριφορά των αγορών. Α περάσω όμω λεπτομέρειες και την ουσία της έκθεσης μου. Ταυτόχρονα όμω, επιτρέψτε μου και να αναφέρω συνοπτικά κάποια από τα συμπεράσματα της έκθεσης. Το 2008 συνετάχθησαν και τι αναλύσει των ε, μεταλλασσομένων δομών στις χρηματοπιστωτικέ αγορές από το 2008 που τώρα φαίνεται ότι προχωρούν σε επαλήθευση, οι χρηματοπιστωτικέ αγορές έχουν ξεφύγει από τα πρότυπα τα στηριζόμενα στις ε, ε τράπεζες ε, προς πρότυπα στηριζόμενα σε διαρθρωμένα χρηματοπιστωτικά συστήματα και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου. Βέβαια αυτό δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι πολλοί από τους ε, οργανισμούς της επιχειρήσης της χώρας σας εξαρτώνται ιδιαίτερα από, την, ε, από το μοντέλο που στηρίζεται στις τράπεζες. Ωστόσο, και, ε, στην, και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και χώρες όπως η Ολλανδία, η Ιρλανδία έχουν στηριχθεί σε μοντέλα, τελευταία τουλάχιστον στηρίζονται σε μοντέλα χρηματοπιστωτικά και στήριξης ασφάλισης των κεφαλαίων. Βέβαια, δεν είναι κακό πράγμα αυτό απαραίτητα, αλλά η εξασφάλιση των κεφαλαίων αποτελεί έναν κίνδυνο που δεν είναι προφανής, δεν ήταν τουλάχιστον εξ αρχής προφανής για τις ρυθμιστικές αρχές και μπορεί να προκαλέσει επιπλέον συστημικό κίνδυνο. Το είδαμε και από τι Ηνωμένε Πολιτείε όπου ο αρχηγός κεντρική τράπεζα, ο πρόεδρος τη Κεντρική Τράπεζα, ο Γκρινσπαν είχε κρίνει ότι δεν μπορεί ένα τέτοιο μοντέλο να προξενήσει συστημικό κίνδυνο, δηλαδή η στήριξη τη ασφάλεια κεφαλαίου, στην ασφάλιση κεφαλαίου μπορούσε να προκαλέσει την επέκταση τη αγορά, να την καταστήσει πιο γερή την αγορά, να την ενισχύσει κτλ. Αλλά ο κίνδυνο με το να αναπτύξουμε συστήματα ασφάλιση σε όλη την αγορά δεν εξαφανίζεται. Σε μικροεπίπεδο επίση, είδαμε ότι ορισμένε Τράπεζε τράπεζες μετακινήθηκαν προς πρότυπα καταρρεμπημένα τα λένε ορισμένοι, εμείς τα λέμε ε, επανεγκατεστημένα μάλλον, που σήμαιναν απλώς μετακίνηση του κινδύνου για να μπορέσουν έτσι να χειριστούν τα ζητήματα, να διατυπώσουν κατά τρόπο πιστικό το ισοζυγιό τους με αποτέλεσμα όμως απλώς να μετακινούν τον κίνδυνο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά τρόπο ιδιαίτερα περίπλοκο, με συνέπεια και αδιαφάνεια στις αγορές και δυσκολία για τις ρυθμιστικές αρχές να επιθεωρούν, να παρακολουθούν τον κίνδυνο και την αδυναμία να μεταβληθεί ο συστημικός κίνδυνος από το κεφαλαιοχικό αυτό σύστημα, το σύστημα εξασφάλισης των κεφαλαίων και μικρότερη προβλεψιμότητα. Δηλαδή, τελικά για να ρυθμιστεί ένα, για να διορθωθεί ένα πρόβλημα, οι διορθωτικέ κινήσει πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερε με τον νέο αυτό πρότυπο. Επίση, πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρχαν πολλές συναλλαγέ και πέραν των συνόρων μέσω τραπεζών και θηγατρικών τους και άρα το πρότυπο του ενό διαβατηρίου όπω ονομαζόταν όπου μπορούσε κανείς να στηριχθεί στον, στη μία εποπτική αρχή για μία τράπεζα και μπορούσε αυτή η εποπτική αρχή να παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές στις τράπεζες, δεν αρκούσε, διότι αυτή η εποπτική αρχή ή δεν είχε κίνητρα ή δεν είχε αρκετές πληροφορίες ή εξουσία για να παρακολουθήσει τις δραστηριότητες της τράπεζας σε άλλο κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τέλει δηλαδή, αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερο συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, κατά κάποιο τρόπο να αναπτύξουμε τη διαδικασία Λαμφαλούση με τις επιτροπές ε, επίπεδου 3 που θα πρέπει να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα ώστε να έχουν και καλύτερη ικανότητα να συντονίζουν σε εποπτικές δραστηριότητες επίπεδο κρατών μελών, όχι να μετατραπούν σε εποπτικές αρχές, αλλά να συντονίζουν τις ε, δραστηριότητες των εποπτικών οργάνων των κρατών μελών. Και επίσης σημαντικό για μας ήταν ότι οι εποπτικές αρχές, οι εθνικές εποπτικές αρχές στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι υπόλογες να υπάρχει ένας λογαριασμός λογοδοσίας όχι μόνο προς το Υπουργείο των Οικονομικών ή την, της Οικονομίας ή του, τη Βουλή αλλά να είναι υπόλογες και προς άλλα κράτη-μέλη εκεί όπου έχουν δραστηριότητε δηλαδή οι εθνικές τους ε, τράπεζες, οι τράπεζες του κράτους μέλους δηλαδή. Άρα να υπάρχει ένα πλέγμα ελέγχου και, και όχι απαραίτητα πολύ ψηλή εναρμόνιση όπως τα πρόβλεπε η ενία ευρωπαϊκή πράξη το 86 που τελικά εκείνη την εποχή είχε νόημα βέβαια αλλά τώρα δεν χρειάζεται. Τώρα χρειάζεται μια αναδιάρθρωση της χρηματοπιστωτικής ε, εποπτείας στην Ευρώπη. Επίσης επικρίνουμε τη Βασιλεία 2. Και πριν από την κρίση το είχαμε πράξει αυτό το 2005 ο Τζον Νίκουελ και εγώ ε, συντάξαμε ένα βιβλίο όπου επικρίναμε απερίφραστα τη Βασιλεία 2 γιατί στηρίζεται μόνο στην μικροπροληπτική εποπτεία, δηλαδή σε τράπεζες των οποίων τα διαχειριστικά πρότυπα είναι μόνο πρότυπα οικονομικά, κεφαλαϊκά, οικονομικά, ενώ ο γενικός στόχος της Βασιλείας 2 βέβαια ήταν καλός, δηλαδή να υπάρχει ένας τρόπος να ενισχυθεί η διαχείριση του κινδύνου για τις ε, τράπεζες, αλλά αυτό ε, μπορεί να ήταν ε, η απειλή, αλλά το κίνητρο στην προκείμενη περίπτωση ήταν ότι εάν ε, μία τράπεζα πιανόταν σε υψηλό επίπεδο κινδύνου θα μπορούσε να μειώσει το ποσοστό ή την ποσότητα κεφαλαίου εποπτείας αντίστοιχα. Είχε λοιπόν αυτό το ελάττωμα το σύστημα της βασιλείας και έπρεπε να διορθωθεί. Αλλά επαναλαμβάνω δεν ήταν αυτός ο λόγος της, πιστο, της κρίσης της χρηματοπιστωτικής είχε να κάνει αυτή περισσότερο με τον κίνδυνο της ρευστότητα που ήταν ήδη εμφανής στην, ε, στη χονδρική κεφαλαιοχική αγορά, όπου πάλι τα κράτη-μέλη έπαιζαν το δικό τους ρόλο, ε, είχαν και αυτά ένα ρόλο δηλαδή να δραματίσουν, αλλά δεν οφειλόταν μόνο σε ένα κράτος, σε μία τράπεζα τα προβλήματα η εξωτερικότητα λοιπόν των κινδύνων, οι υπερσυνοριακές συναλλαγές ε, ε, σημαίνουν ότι θα πρέπει και η νομοθεσία να επιβάλλει υπερσυνοριακή εστίαση, δηλαδή οι εποπτικές αρχές να έχουν πιο γερούς και διαρκείς δεσμούς μεταξύ τους πέραν των συνόρων και να υπάρχει η εποπτεία, η αμοιβαία, ε, με σεβασμό βεβαίως ε, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των ολοκληρωμένων χονδρικών αγορών κεφαλαίων το, η αγορά ανταλλαγής ε, κινδύνου πιστώσεων είναι ένα χαρακτηριστικό αυτής ε, της υπόθεσης. Τώρα θα το δούμε αργότερα. Και έτσι βλέπουμε κάποιους, ε, κάποια ρυθμιστικά και κάποια υποπτικά θέματα ε, Πάλι επαναρχόμαστε Βασιλεία 2 γιατί έχει την επικαιρότητά τη, την ακούμε στα μέσα μαζική ενημέρωση. Μερικέ φορέ μάλιστα ορισμένοι την αποκαλούν και Βασιλεία 3 γιατί έχει σε μεγάλο βαθμό μεταρρυθμιστεί τουλάχιστον από τι ε, πρόσφατε προτάσει τη Επιτροπή τη Βασιλεία. Προτάσει οι οποίε βαίνουν προ την ουσιαστική κατεύθυνση αλλά πάλι είναι ανεπαρκεί και πάντω στηρίζονται σε μια εσφαλμένη ανάλυση. Η πρόταση πάντως τώρα φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη των, τις επιπτώσεις της ανάληψης κινδύνου για το μικροκεφάλαιο και είδαμε ότι υπήρξε αύξηση του ποσοστού ανάρτησης και για πρώτη φορά από τη Βασιλεία και της, του κινδύνου για την ρευστότητα. Δηλαδή για πρώτη φορά συζητήθηκε το σε ποιο βαθμό η χρηματοδότηση μπορεί να στηρίζεται ή πόσο μπορούν να εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση από τις αγορές, τις χονδρικές αγορές κεφαλαίου. Ναι, Ωστόσο δεν νομίζουμε ότι έχει δοθεί αρκετή προσοχή στις ε, μακροοικονομικές επιπτώσεις του πλαισίου της Βασιλείας 2. Και αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, επίσης ασχολούμεθα με ένα σημαντικό θέμα πώς θα, μπορούμε, πώς θα γίνονται οι δοκιμασίες ε, για συνθήκες πίεσης. Και υπάρχει ένα σχετικό θέμα που αφορά τις μεγάλες τράπεζες, τι διαχείρισης, τι είδους μοντέλο διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει να έχουν. Θα πρέπει οι ρυθμιστές να ασχοληθούν με το θέμα αυτό, να προσπαθήσουν να βρουν τρόπους να περιορίσουν τη δυνατότητα μεγάλων τραπεζών ανάληψης κινδύνου στις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτά είναι σημαντικά θέματα και ενδεχομένω θα μπορούσα να πούμε ότι αυτό το οποίο συμπεραίνουμε από, το, από τη ρίση too big to fail, γιατί οι Τράπεζε συνήθω λειτουργούν σε μια ομαδική δομή, σε μια συλλογική δομή. Υπάρχουν διάφορε ξεχωριστέ οντότητε της εταιρείε που, έχουν, που εμπίπτουν σε διάφορα δικαιοδοτικά συστήματα σε διάφορες χώρες του κόσμου. Ε, συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς σε μια τράπεζα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ένα ορισμένο μέγεθος γιατί η τράπεζα έχει διάφορες θηκατρικές που μπορούν να τις ελέγχουν είτε άμεσα είτε έμεσα. Συνεπώς υπάρχει πολύ περιθώριο για αρμπιτράζ. Εμείς αυτό το οποίο λέμε και είπαμε, γιατί είναι πολύπλοκη η διάθεση των τραπεζών, ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε την εφαρμογή μεγαλύτερων φόρων σε σχέση με το μέγεθός τους αλλά με τη διάσταση του κεφαλαίου τους είναι εξωτερικός ε, φόρος. Μας αρέσουν οι μεγάλες τράπεζες αν μπορούν να δημιουργήσουν μεσότερε θέσεις ε, απασχόλησης, να κάνουν περισσότερες επενδύσεις, αλλά ενέχουν συστημικούς κινδύνους. Συνεπώς θέλουμε να εσωτερικεύσουν αυτό το συστημικό κίνδυνο ε, πληρώνοντας ένα υψηλότερο κόστος επειδή έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις, άρα έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία. Συνεπώς λοιπόν είναι μια οικονομικά πιο αποτελεσματική προσέγγιση αντί να έχουμε αυτές τις σχετικά αυθαίρετες, τους αυθαίρετους νομικούς ε, περιορισμούς. Και βεβαίως ε, όσον αφορά τα CDS είχαμε μια άλλη έκθεση στην Επιτροπή ΕΚΟΝ που λέει ότι οι συμβάσει για τα παράγωγα θα πρέπει να διαμορφωθούν στα, στα κέντρα συμψηφισμού ε, και θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα με τις ε, πιστώσεις γιατί το επίπεδο χρέους είναι αυτό το οποίο ε, δημιουργεί τον κίνδυνο για ολόκληρο το σύστημα. Θα πρέπει να λειτουργούν αυτά τα κέντρα συμψηφισμού τα οποία όμω δεν είναι τίποτα άλλο από χρηματοπιστωτικέ οντότητε που δημιουργούνται από τις τράπεζες. Τι πρώτε φορέ οι ιδιοκτήτες είναι τράπεζες. Και ναι, μεν επιτρέπουν περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά του κινδύνους, αλλά δεν ε, ρυθμίζονται από, με μέτρα νομοθετική ε, εποπτείας ε, στην Ευρώπη. Δεν ξέρω. Δεν νομίζουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη ρύθμιση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει μια ρύθμιση εσείς με τα κέντρα συμψηφισμού στις Ηνωμένε Πολιτείε αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι παρέχουν σημαντικά ωφέλη αλλά δεν έχουν ρυθμιστεί για τα κεφάλαια Πρόσφατα ε, ε, δημοσιεύτηκε ένα πολύ καλό άρθρο που έδειξε ένα από αυτά τα κέντρα συμψηφισμού, Ινστιτούτο Συμψηφισμού στο Λονδίνο. Διαμαρτυρήθηκε γιατί ένα βελγικό Ινστιτούτο ε, προσέφερε πολύ χαμηλά περιθώρια για τα ασφάλιστρα κινδύνου και είπαν ότι ήταν παράλογα χαμηλά αυτά τα περιθώρια και δεν ήταν αρκετά για να γίνει διαχείριση του κινδύνου. Νομίζουμε λοιπόν θα πρέπει να διατυπωθούν κάποιε ελάχιστε προδιαγραφέ. Οι ε, ζητήματα εποπτεία θα πρέπει να τεθούν εδώ. Επίση, σημαντικό για την Ευρώπη είναι ο αντίκτυπο των ε, διεθνών ρυθμίσεων όσον αφορά τις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές και οι επιπτώσεις της Βασιλείας 3 ή των θεμάτων μόχλευσης θα έχει μια σημαντική επίπτωση στη, στη χορήγηση δανείων από τις ε, τράπεζες σε πολλά δικαιοδοτικά συστήματα στην Ευρώπη. Ε, και θα υπάρξει ένα δίλημα όσον αφορά την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσει και την εφαρμογή της. Τώρα όσον αφορά τι μεταρρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις, επεξεργαστήκαμε τις ε, προτάσεις της σχετικής έκθεσης στις, στο πλαίσιο συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο και θα υπάρξουν μάλλον κάποιες ε, τροπολογίες όσον αφορά από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, διαχείριση συστημικού κινδύνου. Νομίζουμε ότι είναι ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, γιατί εντάσσει κάποιες παρατηρήσεις από την έκθεση του 2007 Δηλαδή θα πρέπει να παγιωθεί περισσότερο, να εδρεωθεί η εποπτεία στην Ευρώπη των χρηματοπιστωτικών αγορών, αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένα καθεστώς για τα ευρωπαϊκά ψηφίσματα. Ε, αυτό που βασίζεται στην παρούσα οδηγία είναι ανεπαρκές. Έχουμε κάποια προβλήματα σε σχέση με αυτό, την απουσία αποτελεσματικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, όσον αφορά τις διεθνείς ε, προδιαγραφές και τη φορολογία για τις χρηματοπιστωτικές ε, συναλλαγές. Νομίζουμε ότι αυτή η φορολογία είναι πολύ σημαντική ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Ε, τώρα, οι νέες για το Βασιλεία 2 από τον περασμένο Δεκέμβριο πιστεύουμε ότι είναι ανεπαρκή. Γιατί παρόλο που το θέμα διεθνώ είναι το πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μακροοικονομική εποπτεία ε, για να αντικαταστήσει τη μικροοικονομική εποπτεία, νομίζουμε ότι είναι ακόμα ανεπαρκή οι προτάσεις αυτές πλαισίωσης. Ε, στην έκθεση νομίζω μπορείτε να δείτε καλύτερα. Έχουμε συλλέξει τα δεδομένα από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ευρώπη. Στη δεξιά στήλη έχουμε την αναλογία ε, μόχλευσης που έχουν αυτές οι τράπεζες οι τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν αυτές τις αναλογίες μόχλευσης. Είναι η αναλογία μετοχών ε, ε προς κεφάλαια, προς διαθέσιμα. Ε, υπάρχουν τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν υψηλότερες αναλογίες μόχλευσης, κάτι το οποίο είναι καλό. Αλλά στην Ευρώπη είναι οι αναλογίες αυτές πολύ χαμηλότερες. Είναι συγκρίσιμη η αριθμή αυτή ε, μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής ή θα μας οδηγήσουν σε διαφορετικά συμπεράσματα σχέση με το σύνολο των διαθεσίμων. Ε, δεν ξέρω, ε, Ίσως συνάδελφο μπορεί να σα απαντήσει. Θα βάλουμε σε μια υποσημείωση, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Η τυποποίηση των δεδομένων είναι ένα σημαντικό θέμα. Λοιπόν, έχει γίνει μια σχετική μελέτη με σύγκριση ευρωπαϊκών, ε, αμερικανικών και καναδικών τραπεζών σε σχέση με τις ευρωπαϊκές. Πόσο θα έχει η αύξηση της αναλογίας μόχλης, πώς θα επηρεάσει τις τράπεζες στην Ευρώπη στο Διεθνές Νομισματικό, ε, νομίζω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χρησιμοποιεί παρόμοια δεδομένα και έχουν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα. Έχω ένα άλλο, μια άλλη διαφάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο εκπώνησε μια έκθεση πριν από μερικούς μήνες, αλλά δεν ασχολούνται με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Δεν ξέρω. Ε, ίσα μπορούσαν να μας φωτίσει από τους συγγραφείς είναι οι συνολικές ε, κεφαλαϊκές ε, απαιτήσεις. Και αυτό το οποίο συμπεραίνει το IMF είναι ότι στη δεξιά στήλη βλέπουμε ε, τις ευρωπαϊκές τράπεζες και τα χρήματα που απαιτούνται για να είναι συμβατές με, το, με την απαιτούμενη αναλογία μόχλευσης. Η άλλη στήλη είναι οι τράπεζες στο Ηνωμένο που θα πρέπει να έχουν χαμηλότερα επίπεδα κεφαλαικών απαιτήσεων ε, για να συμφωνήσουν με τα επίπεδα μόχλευσης, με την αναλογία μόχλευσης που ορίζει η Βασιλεία ενώ οι τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να έχουν κάπως ε, περισσότερα χρήματα, περισσότερα κεφάλαια. Τώρα, αν δούμε τη δεύτερη στήλη, αυτό είναι το καλύτερο, το ποιότητας κεφάλαιο ως αναλογία κινδύνου προς διαθέσιμα. Η Επιτροπή Βασιλείας είπε ότι η αναλογία θα πρέπει να είναι 10%. 8% ήταν στο Βασιλεία 1 και 10% θα πρέπει να είναι στο Βασιλεία, ε, προβλέπει Βασιλεία 2. Αυτό θα ήταν πιο δύσκολο στι Ευρωπαϊκέ Τράπεζε, γιατί θα πρέπει να έχουν 380 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια για να συμφωνήσουν με το 10% αναλογία, ενώ οι Βρετανικές τράπεζες πολύ λιγότερα. Γιατί, Γιατί οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί, Ευρωπαίοι επόπτες έχουν would classify as Έχουν μετοχές που είναι επιβαρημένες με χρέος. Και έτσι αξιολογούνται, αξινομούνται. Συνεπώς, η νέα πρόταση της Βασιλείας είναι αυτή η ταξινόμηση για τα κεφάλαια που επιβαρύνονται με χρέο. Λοιπόν, άρα γίνεται πιο συμμορφώνεται με το 10%. 8% πάμε στη Βασιλεία 1. Βλέπετε οι ευρωπαϊκές τράπεζες ε, δεν τα πανάσχε με το 8%. Θα έπρεπε να θεωρήσουν ότι το κεφάλαιό του σε επίπεδο είναι απλέ μετοχέ και το ποσοστό του είναι 150 δισεκατομμύρια. Αλλά το κόστο του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Αμερική είναι λιγότερο, διότι προσχω... συμμορφώθηκαν περισσότερα με τι κοινέ μετοχέ, που είναι το κύριο μερίδιο του κεφαλαίου κατηγορία 1. Οπότε για να περάσουν στην κατηγορία Βασιλεία 2 θα έχουν μικρότερα προβλήματα από τι Ευρωπαϊκέ Τράπεζε. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα αυτή, αυτό το διάγραμμα δείχνει το Federal Reserve με στοιχεία για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη ΣΥΠΑ, αλλά όχι για την υπηρετική Ευρώπη. Εξετάζει το θέμα του κατά πόσο στοιχεία ενεργητικού είναι σε τίτλους και ποια δεν είναι. Και βλέπουμε το πρώτο τρίμηνο του 2009, παρόλο που υπήρχε η, κρίση και ήταν πιο περιορισμένο ε, η έκδοση τίτλων, βλέπουμε οι τράπεζε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν περίπου 60% του στοιχείου ενεργητικού σε αξιόγραφα και σε δάνεια για, σε νοικοκυριά και για στεγαστικά δάνεια. Στη δεξιά στήλη το πρώτο τρίμηνο του 2009 και τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού. Τα περισσότερα στοιχεία ενεργητικού εξακολουθούν να εκδίδονται από Αμερικανικέ και Βρετανικέ τράπεζε υπό τη μορφή τίτλων. Και αυτό είναι καλό, διότι παίρνει ρευστότητα όταν το κάνει αυτό. Ε, οπότε μπορεί να ελέγξει τον κίνδυνο. Ε, τώρα, τιτλοποίηση σε χαμηλότερο επίπεδο στη ΣΥΠΑ και στη Βρετανία και πιστοτικές κάρτες και στεγαστικά βλέπετε πολύ χαμηλότερο επίπεδο έκθεση τίτλων. Ε, δεν είναι ε, χρέο, αλλά ε, η τιτλοποίηση εξακολουθεί να είναι κάτι ζωντανό, να κινείται και να ζωντανεύει την οικονομία. Δεν θέλουμε να το σκοτώσουμε, θέλουμε να το ελέγξουμε καλύτερα για να μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερου κινδύνου. Τώρα πιο γρήγορα απλώ να αναφερθώ στα λάθη όσον αφορά τη των κινδύνων. Ένα από τα προβλήματα με τα μοντέλα τη διαχείριση του κινδύνου, ποιο ήταν ότι τα μοντέλα διαχειρίσεως του κινδύνου υποτιμούσαν τον κίνδυνο ε, που, ε, που βασιζόταν σε εσωτερικά στοιχεία που αφορούσαν την τράπεζα για να κάνουν την πρόβλεψη. Έβλεπαν τι γινόταν στον τομέα της συγκεκριμένη τράπεζας, πιθανότητα ε, μη τήρησης των υποχρεώσεων σε διάφορες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, ε, και εξετάζουν τα στοιχεία για περιορισμένο χρονικό διάστημα, κανονικά δεν λαμβάνουν υπόψη τι συνέπειε ε, μια κρίση ρευστότητα ή ενό πομφόλιγα που εκρήγνεται και βασίζονται στο μοντέλο του. Αυτά είναι μοντέλα που είναι καλά για κανονικέ εποχέ και όχι προβληματικέ. και επίση τα μοντέλα δεν κάνουν μακροοικονομικούς συσχετισμούς, ε, δεν λαμβάνουν υπόψη επενδυτική συμπεριφορά που είναι εκτός της τράπεζας αν αποφασίσουν ε, όλοι, τα, όλοι οι καταναλωτές, ε, οι επενδυτές να μην αγοράσουν τα χρεόγραφα της τράπεζας. Τι γίνεται. Βλέπουμε λειτουργικό κίνδυνο, ε, επιχειρηματικό ρίσκο και όχι κίνδυνο ρευστότητα. Αγνοούν τον κίνδυνο ρευστότητα που είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Οπότε τα μοντέλα θα πρέπει να αναδιαθωθούν. Τα μοντέλα για να λάβουν υπόψη μακροστοιχεία όσον αφορά τη συνετή διαχείριση. Τώρα αναφερθώ στο, στην Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Συστημικό Κίνδυνο. Μιλήσαμε για το Ευρωπαϊκό Σύστημα τη Δημοσιονομική Εποπτείας και την το e SRB είναι αυτό το, το, η Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου είναι κάτι καλό για μακροοικονομική μακροοικονομικό έλεγχο συνετής διαχείρισης. Η Ευρώπη έκανε εποπτή σε επίπεδο μικροοικονομικό. Αυτός ο φορέας θα δηματίσει σημαντικό ρόλο. Υπάρχει νομικό θέμα για το πόσο ε, ποια είναι η νομική βάση, είναι το 114 τη συνθήκη τη Αβώνα, θέμα υπείου δικαίου. Είναι η νομική βάση επί την οποία χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δημιουργήσει αυτή την επιτροπή του συστημικού κινδύνου. Ε, και υπάρχει κάποια ανησυχία από κάποιου νομικού ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και από πλευρά άλλων νομικών υπάρχουν ανησυχίε ότι αυτή η Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου δεν έχει ορθή νομική βάση σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις αργότερα αλλά ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτό ισχύει είναι διότι οι οικονομολόγοι δεν καθορίζουν συστημικό κινδύνο επαρκώς, ξεκάθαρα. Όλος σκοπός της ύπαρξης της Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου είναι να παρακολουθούν για μακροοικονομικούς λόγους το συστημικό κίνδυνο. Πρέπει να ξέρει τι είναι συστημικός κίνδυνος για να κάνει την εποπτεία. Και αυτό είναι για να έχει ασφάλεια δικαίου στον ορισμό όσον αφορά την ε, εξουσία που έχει αυτό ο φορέας. Υπάρχει συζήτηση μεταξύ των, νομικών, ε, ποιος είναι των οικονομολόγων είναι συστημικός κίνδυνος. Άρα ο δικαστής μπορεί να πει ότι δεν έχουμε σαφή ορισμό του συστημικού κινδύνου. Οπότε μακροοικονομική εποπτεία συνετής διαχείρισης. Τώρα ο κανόνας Βόλκερ είναι εξέλιξη στη ΣΥΠΑ αυτή. Ε, η ύπα δεν προτείνει ε, να αλλάξει τα πάντα, αλλά θέτει περιορισμούς αφορά τις τράπεζες που έχουν ασφαλείς αποταμιεύσεις δεν μπορούν να επενδύσουν σε hedge funds και σε ιδιωτικά χρεόγραφα. Αυτό ίσως να είναι καλό για τη ΣΥΠΑ και όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό στις απαντήσεις θα το ξεκαθαρίσω. Χρειαζόμαστε ολιστική προσέγγιση, σφαιρική προσέγγιση στη ρύθμιση, πιο απαλές κεφαλουχικές απαιτήσει και ρευστότητα, ε, τι γίνεται σε διασυνοριακό επίπεδο και θα πρέπει το τραπεζικό σύστημα να βασίζεται περισσότερο σε διαχείριση συστημικού κινδύνου και όχι σε χρηματοδότηση σε χοντρικό επίπεδο. Και μετά όσον αφορά τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα τον αναλύσω αργότερα. Ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο ε, είναι διστακτικό όσον αφορά το φόρο αυτό για τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ. Αλλά αν το επίπεδο είναι χαμηλό των φόρων δεν θα υπάρχει στρέβλωση τη αγορά μεγάλη και γι' αυτό ο φόρο αυτό είναι σημαντικό των συναλλαγών, των χρηματοπιστωτικών, διότι προσμετρά ε, αντικυκλικής ρυθμίσης. Οι φόροι αυτοί λοιπόν μπορούν να είναι σημαντικό εργαλείο για αντικυκλική ρύθμιση. Οπότε όταν τράπεζες βγάζουν κέρδη και έχουν μεγάλα κέρδη σαν στοιχεία ενεργητικού ε, πληρώνουν πολύ μικρό ποσοστό αυτού του κέρδους σαν φόρο όχι απαραίτητα διότι προσπαθούμε να μαζέψουμε περισσότερα χρήματα για να τροφοδοτήσουμε το έλλειμμα, διότι θέλουμε να μειώσουμε ε, την ανάληψη κινδύνου από την τράπεζα. Διότι αν χρηκοποιήσει η τράπεζα, πολύ συχνά φορολογούμενο πληρώνει το λογαριασμό και τα σπασμένα. Άρα ε, εδώ υπάρχει ρόλο για τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ και στι ρυθμίσει θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την υπομονή σα. Ευχαριστώ. Εκτιμώ την παρουσίασή σα, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα καλώ του συναδέλφου ε, να υποβάλουν ερωτήσει. Έχω την εισηγήτρια που θα είναι πρώτη και μετά θα ακολουθήσουν οι επόμενοι ε, συνάδελφοι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Ήταν πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα και διαφημιστική. Ίσως ήταν σκόπιμο να επισημανθεί ότι η υποτίμηση των συστημάτων ιστορικής ήταν το κύριο πρόβλημα. Και νομίζω ότι αυτά ήταν τα στοιχεία έχουμε δει ήδη στο κοινοβούλιο, για τα οποία έχουμε σαφή συνέντευξη. Δεν θέλω πάντω να ρωτήσω τι έχετε να πείτε για την ε, Επιτροπή τη Βασιλείας, γιατί παραμένει σημείο αναφορά σήμερα. Γιατί <laughs> τη των τραπεζών. Είπατε ότι θα, θα πρέπει, ότι θα πρέπει να έχει μια ολιστική προσέγγιση. Είναι χώρος <laughs> θεμητός για αυτή την ε, ολιστική προσέγγιση η Επιτροπή της Βασιλεία. Έχω και εγώ τι εμφολίες μου. Καταρχά, διότι ό,τι και να γίνει εκεί, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν πρέπει να το εφαρμόσουν και μόνο λένε ότι θα γίνει με τη Βασιλεία 3, χωρί να έχουν ε, επικυρώσει τη Βασιλεία 2. Ενώ εκείνοι ξεκίνησαν τη διαδικασία, προκάλεσαν τη διαδικασία για τη θέσπιση τη και επιπλέον διότι ο μηχανισμό στον οποίο αναφέρεστε, ο οποίο έχει διαδραματίσει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο σε τελευταία ανάλυση στην ε, ή μη τι άλλο επέκταση τη κρίση, η ιστορική φυσιολογία των μοντέλων. Επνέτη, πιστεύω, σε μεγάλο βαθμό από τις μεγάλες τράπεζες επενδύσεων που ανήκουν στις ΗΠΑ ακριβώς. Και άρα ή μη τι άλλο υπάρχει ζήτημα συγκρούσεων συμφερόντων, προφανές, προφανές, προφανές συμπέρασμα. Ένα άλλο θέμα διαφωνία του προ την Επιτροπή τη Βασιλεία είναι παραγωγή γνωρίζω ότι υπάρχουν και μεγάλα σοφά μυαλά εκεί πέρα κτλ και ότι, και άλλωστε και εσείς είστε παράδειγμα αυτού, ότι διαπιστώνουμε ότι τα πάντα βρίσκονται επιτάπητος, όλα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, αλλά μη μας μιλήσετε για συστημικούς κινδύνους. Μη μας μιλήσετε για το too big to fail. Εγώ να σας πω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι πώς μπορούμε να έχουμε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα, ένα τραπεζικό σύστημα, το οποίο να επιτρέπει να λειτουργήσει η πραγματική οικονομία, να επιτρέψει στις τράπεζες να κάνουν τη δουλειά τους. Θα μου πείτε ναι, προϋπόθεση για να κάνουν τη δουλειά τους καλά είναι να μην είναι εκτεθειμένοι σε συστημικούς κινδύνους. Έστω. Αλλά πάλι δεν με πείθει το επιχείρημα. Και θα έλεγα ότι... γιατί, γιατί, γιατί άπαξ και επεξεργαστεί ένα κανόνα η Βασιλεία. Καθόμαστε και το ψάχνουμε δεξιά και αριστερά, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις τα λοιπά και είχαμε κάνει αυτή την ιστορία με τις, ε, με τις ε, επενδύσεις. Αλλά εν τέλει η ισορροπία του κειμένου, τα εσωτερικευμένα, ιστορικευμένοι κίνδυνοι, όλα αυτά τελικά δεν λαμβάνονται και πολύ υπόψη. Σας μιλήσατε για την ελληπή δουλειά της Επιτροπής 3, επίπεδο 3. Ναι, έστω. Αλλά μήπως θα έπρεπε να προχωρήσουμε. Θέλει μια εξέλιξη αυτή η κατάσταση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το μωρό άρχισε να πουσουλάει σιγά σιγά. Οι τρεις επιτροπές επέδου 3 έχουν πιστεύω πια ξεκινήσει τη δουλειά τους, είναι ενωμένε πια. Από την άλλη μας δεν υπάρχει νομική βάση, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τον συστημικό κίνδυνο και στην αρχή είπατε ότι κάτι τέτοιο στον Ηνωμένο Βασίλειο είχε διαφορετική αντιμετώπιση για τους γνωστούς λόγους. Μα το πρόβλημα δεν είναι ο συστημικός κίνδυνος. Το πρόβλημα μεταξύ άλλων είναι η μακροοικονομική επιτήρηση. Πριν να επισέλθουμε στο συστημικό κίνδυνο. Γνωρίζω ποια είναι τα νομικά επιχειρήματα, ξέρω πόσο μπορεί να επηρεάσουν ε, το, τη συζήτηση ενός προβλήματος όπως αυτό της κρίσης της Ελλάδας. Αλλά ένα πράγμα που μπορούμε να αποκομίσουμε σαν δίδαγμα από όλη αυτή την κρίση, και το είπατε και ο ίδιος, είναι ότι η μακροεπιτήρηση είναι ένα ζήτημα κριτικό, ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί σοβαρά. Και ναι, το συζητήσε σε όλος ο κόσμος. Και οι Βρετανοί εμπειρογνώμονες της ομάδας του Ζακ Και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει με αίσθηση ευθύνης να μην ε, διαχέουμε σφαλμένες εντυπώσεις λόγω στην τεχνομική βάση. Το Κοινοβούλιο θέλει να ξαναγυρίσει την αρχική πρόταση της ε, Επιτροπής Λαγοζιέχ, που την υποστήριξε η Επιτροπή και από τη διέλυσε το Συμβούλιο. Εγώ σε αυτό υποστηρίζω στεναρά τη θέση του Κοινοβουλίου. Για δε την ε, αντιστάθμιση. Τα πεδία αντιστάθμισης για τα παράγωγα πιστώσεων τι είδους αρχιτεκτονική προβλέπετε γι' αυτά. Είχαμε κάποιες εταιρείε απόψεων στις ΗΠΑ, ε, αρκετά έντονες θα έλεγα μας με τον Πρόεδρο. Και βέβαια θα πρέπει να αποφευχθεί η, ο, ο πολλαπλωσιασμός ε, των ε, πεδίων αντιστάθμισης. Ευχαριστώ πολύ σημαντικές παρατηρήσεις σας. Ένα σημαντικό τμήμα του Πιλάνα 2, του πλαισίου Βασιλεία 2, δεν αναπτύχθηκε επαρκώ πριν από την κρίση και τώρα είναι μια δυνατότητα να γίνει ακριβώς αυτό και είναι μεγάλη δυνατότητα εκείνη διαμορφώνουν ευρωπαϊκή πολιτική να καλύψουν το κενό, διότι δεν νομίζω ότι υπάρχει σαφής κατανόηση από πλευράς στη Επιτροπή της Βασιλείας τι θα πρέπει να κάνουν οι υποπτικοί φορείς στον πυλώνα 2 εστιάζεται πολύ το πράγμα στα, ε, στον πυλώνα 1, διαχείριση των στοιχείων των τραπεζών, διαχείριση του κινδύνου κλπ. Μοντέλο κινδύνου. Και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά όσον αφορά το δεύτερο πυλώνα, θα πρέπει να σκεφτούμε στην Ευρώπη το πώ ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πρότυπα, ποια κριτήρια, ποια πρότυπα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, οι ρυθμιστικοί φορεί για να καθορίσουμε το πόσο καλό είναι το μοντέλο τη τράπεζα για τη διαχείριση του κινδύνου. Πόσο στέρεο είναι. Αυτό το, αυτά τα μοντέλα για τι μεγάλες τράπεζες είναι κοινά. Χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία όπω είπε, εντό εισαγωγικών για τη του Δεν διαφέρουν αυτά από τράπεζα σε τράπεζα. Τώρα πώς χειρίζονται τα στοιχεία τους, πώ οικοδομούν το μοντέλο τους για επιχειρησιακό κίνδυνο, κίνδυνο αγορά κλπ. Τι δεν λαμβάνουν υπόψη. Δεν λαμβάνουν υπόψη του εξωτερικού παράγοντε. Το πώ εξωτερικοί παράγοντε, το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει το μοντέλο του. Βλέπουν απλώ ότι αν έχουν κάποιες μη ανταποκρίσεις υποχρεώσεις έχουν κάποια στοιχεία ενεργητικού, υποθέτοντας ότι όλες οι τράπεζες θα τα πάνε καλά, ότι άλλες τράπεζες θα είναι εκεί για να αγοράσουν τα στοιχεία ενεργητικού τους. Αλλά τα μοντέλα δεν υποθέτουν τι γίνεται αν όλες οι τράπεζες μαζί δεν μπορούν να βρουν αγοραστή για τα στοιχεία ενεργητικού τους. Όταν το μοντέλο τους λέει ότι πρέπει να πουλήσουν ε, στοιχεία ενεργητικού και αυτό είναι από τα προβλήματα. Τα μοντέλα δεν λάβουν υπόψη την αλληλεξάρτηση, τι αλληλεξαρτήσεις που υπάρχουν όσον αφορά τον κίνδυνο μεταξύ χρηματοσυντικών οργανισμών. Κοιτούν απλώς τον κίνδυνο της τράπεζας εσωτερικά. Ανεξάρτητα από τον εξωτερικό μακρό χρηματοσυντικό τομέα. Και αυτό αφορά τον πυλώνα 2. Η EBA μπορούσε να αναπτύξει αυτό. Συσχετισμό διαχείριση κινδύνου σε ευρύτερα μακροδιαχειριστικά στοιχεία. Λαμβάνοντα επίση συσχετισμού Δηλαδή πώς οι επενδυτές, οι θεσμικοί επενδυτές δρούν σε όλη την αγορά, σε όλη τη χρηματοδοτική αγορά χοντρικής. και εκεί χρειάζονται δοκιμές αντοχής, stress test. Πρέπει να έχεις δοκιμές αντοχής που θα πρέπει να είναι κοινά. Οι τράπεζες τώρα, οι θυμιστικές αρχές πάνε στις τράπεζες και λένε καλώς, τι γίνεται να συμβεί το ένα ή συμβαίνει το άλλο και κάνουν πολεμικό παιχνίδι, πολεμικές ασκήσεις. Θα έπρεπε να λένε τι γίνεται αν όλες οι τράπεζες έχουν το ίδιο πρόβλημα ταυτόχρονα σε όλο το χρηματοδοτικό σύστημα ε, και δεν το κάνουν οι παρούσε δοκιμέ αντοχή. Και αυτό είναι θέμα πυλώνα 2. Γι' αυτό, πυλώνα 2. Κυρία Μπερέ, θυμήθηκα ότι στο σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω τη Ευρωζώνης είχαμε τέτοιο stress test στο υπόμνημα ε, συνεννόησης μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας και το αποτέλεσμα αυτού του μνημονίου που υπεγράφει τον Απρίλιο του 2005 είναι ότι έγιναν οι δοκιμές αντοχής και δεν ανακοινώθηκε ξεκάθαρα στο κοινό το αποτέλεσμα γιατί ήταν φρικτά τα αποτελέσματα. Έγινε stress test δοκιμή αντοχής και αφορούσε όλο το δίκτυο, αλλά τα αποτελέσματα ήταν ικτρά. Α, περισσότερα, απάντηση, περισσότερα πρέπει να, από αυτά πρέπει να γίνουν πιο διαφανή. Μπορεί να τρομάξει η αγορά, αλλά χρειάζεται καλύτερο διάλογο μεταξύ εκείνων που διαμορφώνουν την πολιτική και των θεσμιστικών φορέων. Νομίζω ότι το επενδυτικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει καλύτερα για το πώ οι τράπεζε μπορούν να αντιμετωπίσουν καταστάσει κατά τι οποίε η αγορά αντιμετωπίζει προβλήματα και πιέσει. Στον πυλώνα 2 έχουμε σημαντικό τομέα και χρειάζεται πάρα πολύ ανάπτυξη ρύθμιση σε αυτόν τον τομέα και εκεί μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δραματίσει σημαντικό ρόλο, διότι η Επιτροπή τη Βασιλεία δεν έχει καλύψει αυτόν τον τεράστιο τομέα. οσδήποτε λεπτομέρειε έχουν νόημα, εκτό από αρχέ, καλή διακυβέρνηση κλπ. Μεγαλόσχημων δηλώσεων. Και όσον αφορά την, τον έλεγχο των επιχειρήσεων και τη διαχείριση των επιχειρήσεων, πολλοί διοικητικά συμβούλια τραπεζών έχουν ε, μια επιτροπή κινδύνου και άλλε επιτροπέ οι άλλες κάνουν διαχωρισμό. Οι άλλες, η κάθε επιτροπή έχει ε, δικό τους. Η Επιτροπή Κινδύνου θα πρέπει να έχει άλλα καθήκοντα και ο ελεκτικός φορέας πρέπει να εξετάζει τι κάνει η Επιτροπή Διαχείρισης του Κινδύνου. Και θα έπρεπε στην Επιτροπή αυτή να γίνονται κάποια στοιχεία ενεργητικού και να του πούνε επενδύστε στην αγορά και να προσπαθούσαν να μειώσουν την έκθεσή του και να δουν κατά πόσο θα τα καταφέρουν καλά. Και αυτό θα κάνει αυτέ τι επιτροπέ να συμμετέχουν περισσότερο με αυτά που, σε αυτά που κάνουν οι χειριστές του κινδύνου σε επίπεδο μεσαίο στην τράπεζα. Υπάρχει απομάκρυνση από τις πλευράς επιτροπών διαχείρισης κινδύνου σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου. Πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο ε, σε δοκιμές. Η τράπεζα θα έπρεπε να τους δίνει ένα χαρτζιλίκι και να τους πει «Κάντε το δικό σας χαρτοφυλάκιο, να δούμε τι θα κάνετε». Ε, αυτά σχετίζονται με τον πυλώνα 2 όλα αυτά και νομίζω ότι η ίδια η δίκηση της τράπεζας θα πρέπει να αναδιαθρωθεί αλλά θα πρέπει να αναδιαθρωθεί σε συνεργασία με τον υποπτικό φορέα ε, ούτως ώστε όλοι αυτοί οι κίνδυνοι να αναγνωριστούν, να ανοιχνευτούν και να ελεγχθούν τέλος η Επιτροπή της Βασίλειας, συμφωνώ γιατί θα έπρεπε η Ευρώπη να περιμένει για την Επιτροπή της Βασιλείας να αποφασίσει τι θα κάνει. Η Ευρώπη βεβαίως πολλές από τι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσης είναι μέλη της, Επιτροπή τη Βασιλεία, αλλά η Ευρώπη μπορεί να έχει το πλεονέκτημα του να κινηθεί πρώτη, να είναι δραστήρια, να τροποποιεί την οδηγία για τα κεφαλαιοχικέ απαιτήσει, να ξεκινά ένα διάλογο με την EBA, την Ευρωπαϊκή Αρχή για τι Να πει α κάνουμε αυτό με τον πυλώνα 2, α αναδιαθρώσουμε τη διαχείριση του κινδύνου. Και να μην περιμένουμε για την Επιτροπή τη Βασιλεία και του Αμερικανού να συμφωνήσουν και του Ιαπωνέζου να συμφωνήσουν. Και τότε η Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει την Επιτροπή της Βασιλείας. Και τότε μπορείτε να πείτε για το λόγο προς όφελος των παγκοσμίων συνθήκων για, για το καλό της παγκόσμιας αγοράς κάντε το κι εσείς και να μην είναι τόσο παθητική η Ευρώπη. Και ε, αυτό με ανησυχούσε πάντα όσον αφορά το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάντα είχαμε το συνέστημα ότι πρέπει ε, να μην, να μην προσπαθούμε να κάνουμε πολλά στι Βρυξέλλε, γιατί ασχολείται με αυτό η Επιτροπή τη Βασιλεία και άλλοι διεθνεί φορεί. Και είχαν λόγο να το κάνουν αυτό, διότι ιστορικό πώ επί μακρόν το Ηνωμένο Βασίλειο δραμάτισε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην Επιτροπή τη Βασιλεία και η Επιτροπή τη Βασιλεία έκανε πάρα πολλά καλά πράγματα για τη ρύθμιση των τραπεζών. Όμω ε, κάνανε και κάποια λάθη. Και η Βασιλεία δίνει ένα παράδειγμα ότι το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο καλό. Άρα χρειάζεται να έχουμε ένα μείγμα μεταξύ αυτών που συμβαίνουν σε επίπεδο Επιτροπή Βασιλεία και η Ευρώπη από την άλλη να κινείται. Και οι δραστηριότητε τη Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και οι άλλοι, όλοι μπορούν να σημαντικό ρόλο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω και να επηρεάζουν τα πρότυπα και μετά αυτά να διαβιβάζονται σε επίπεδο τη Επιτροπή τη Βασιλεία. Καλώ, λέει ο Πρόεδρο. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Στην πρωινή συνεδρίαση αυτή τη Επιτροπής εγώ παρουσίασα ένα θεματικό έγγραφο και οδηγήθηκα στα συμπέρασμα ότι οι χρηματοπιστωτικέ και αρχέ αρχές εμπιστεύονται υπερβολικά τα μαθηματικά μοντέλα. Σε μια κρίση παρατηρούμε μια νοοτροπία είναι δύσκολο να έχουμε ένα μοντέλο το οποίο να αντανακλά την πραγματική κατάσταση. Τέλος, μια κρίση είναι ένα καταληκτικό γεγονός της, ε, μέσα σε μια αγορά και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί βασίζονται στα ίδια μοντέλα για να δοκιμάσουν την ε, ρευστότητα στην αγορά. Τα δικά μου συμπεράσματα δεν ήταν να επιβληθεί φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά θα ήταν τιμωρητικό, τιμωρητικό κάτι τέτοιο. Οι δικές μου συστάσεις ήταν τέσσερις και δεν ξέρω κατά πώς θα θέλετε να τις σχολιάσετε. Υπάρχουν τέσσερα σημεία και θα πρέπει να τα διαβάσω. The first one was to... Πρώτο αφορούσε να αυξηθεί το κεφάλαιο ε, σε εταιρείε ε, χωρίς να βασίζεται κανείς σε μαθηματικά μοντέλα. Να υπολογιστεί έκθεση σε ρίσκο για να αναγνωριστεί ο κίνδυνος ε, έκθεση σε σταθείς συνθήκες της αγοράς. Ένα προβλέψεις που να βασίζεται σε διαφορετικούς δείκτες. Και γιατί ένα από τα προβλήματα που αφορά τα παράγωγα είναι ότι δεν είναι για αρκετό χρόνο στην αγορά ώστε να μπορέσει να αξιολογήσει κανείς την αποδοτικότητα, της του ως προϊόντα. Δεν έχουμε δυνατότητα επαρκών προβλέψεων. Ναι, ασφαλώς χρειαζόμαστε αύξηση κεφαλαίου στο ενεργητικό. Ε, εννοείται τιτλοποιημένα διαθέσιμα. Δεν ξέρω. Το θέμα εδώ είναι ότι όταν δεν υπάρχει ρευστότητα, μπορεί κανείς να βασιστεί στα μαθηματικά μοντέλα για μια αξιολόγηση. Εάν δεν μπορεί να γίνει αυτή η αξιολόγηση, θα πρέπει, κανείς, θα πρέπει να μπορεί να κρατηθεί το κεφάλαιο. Νομίζω ότι ο κίνδυνος ρευστότητας είναι κάτι που αντιμετωπίζουν όλα τα ενεργητικά σε κάποιο βαθμό και είναι δύσκολο να υπάρξουν κεφαλικές απαιτήσει. Ε, αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι ότι οι τράπεζες μπορούν να πάρουν τα κεφάλαιά τους, να τα βγάλουν από το φύλλο και να πούν ότι δεν υπάρχει κανένας ε, κίνδυνος, δεν χρειάζεται να κρατήσουμε το κεφάλαιο. Ο ε, το, το ρίσκο μετατοπίστηκε στους επενδυτές που ξέρουν να τον ε, διαχειριστούν, θεσμικοί επενδυτές. Και οι τράπεζες πίστεψαν ότι με το ροφό ξεφορτώθηκαν το κίνδυνο, αλλά ο κίνδυνος ήταν εντός του συστήματος και μόνο το γεγονός ότι τιτλοποιήθηκε δεν σημαίνει ότι απαλλάχθηκαν από τον κίνδυνο. Γι' αυτό οι μακροοικονομικές, η μακροοικονομική υποπτή είναι πιο σημαντική. Θα πρέπει να έχουμε, συμφωνώ μαζί σας, κεφάλαιο το οποίο συνδέεται με το κίνδυνο ο οποίος έχει δημιουργηθεί μέσα στο σύστημα. Αυτό είναι σημαντικό. Όχι τόσο να συνδέεται μαθηματικά μοντέλα, αλλά το γεγονό ότι συνδέεται με μαθηματικά μοντέλα, αλλά ο κίνδυνο υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει και δεν θα πρέπει να δίνουμε τέτοια σημασία στα μαθηματικά μοντέλα. Η εκπόνηση μοντέλων είναι εντάξει, συνδέεται με τη θεωρητική σκέψη. Ε, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε αυτά τα μοντέλα. Βασιλεία, διαστηρίζετε σε τέτοια μοντέλα. Αλλά τα μοντέλα μέχρι, τότε, μέχρι τώρα υπερβολικά σε ιστορικά δεδομένα και δεν έλαβαν υπόψη τους το, τον τύπο των σοκ που είχαμε στην παρούσα κρίση. Νομίζω ότι η υπερβολική εμπιστοσύνη στα μαθηματικά μοντέλα όντως είναι επικίνδυνη. Θα πρέπει να έχουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση στην εξολόγηση των κινδύνων. Νομίζω ότι όλες οι προτάσεις σας είναι πολύ σημαντικές γιατί περιλαμβάνουν υψηλότερο κεφάλαιο. Χρειαζόμαστε περισσότερα κεφάλαια ε, σε μακροβάση, γιατί ο κίνδυνος ενυπάρχει στο σύστημα. και στο τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να ελέγχουμε την υπερβολική άνοδο των τιμών των κεφαλαίων. Στην, στο Βασίλιο Βασίλειο στο παρελθόν είχαν οι τράπεζες δεν είχαν έλεγχο επί των δανείων που χορηγούσαν. Ε, είχαν, ποιοτικό έλεγχο στα δάνεια ε, στο παρελθόν. Ε, ενδεχομένως θα πρέπει να επανέλθουμε σε ένα τέτοιο είδο ε, ποιοτικού ελέγχου. Γιατί αν θέλουμε να έχουμε μακροεπιτήρηση για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί θα πρέπει να παρακολουθούμε τον κίνδυνο. θα πρέπει να συνδέσουμε την αύξηση των τιμών με τον κίνδυνο. Αλλά βεβαίως το περισσότερο, η αύξηση του κεφαλαίου είναι σημαντική. Αλλά πώς ε, μπορείτε να το ορίσετε στην Ευρώπη, στην ε, Μεγάλη Βρετανία ε, και στην Αμερική έκαναν ένα τέτοιο ορισμό. ως μετοχές σχετικές επενδύσεις. Νομίζω ότι αυτό συνεπάγεται ένα μεγαλύτερο κόστος προσαρμογής για τις ευρωπαϊκές τράπεζες από ό,τι για τις αμερικανικές τράπεζες, τράπεζες της Μεγάλης Βρετανίας, που βεβαίως είναι επίσης ευρωπαϊκές, αλλά εμπίπτουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Νομίζω όμως ότι αυτά τα σημεία ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Όλε Σμιτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω κύριο Σμιτ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Κάποιε ερωτήσει και σχόλια. Ξεκινώντα, είπατε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι δραστήρια αυτό εξυπακούεται. Αλλά σε παγκοσμιοποιημένο κόσμο είναι καλό να είσαι και παγκόσμιο σε εμβέλεια και να μην πηγαίνει πολύ γρήγορα. Διαφορετικά κινδυνεύει να μείνει πίσω μόνο και έρημο. Και πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Διαφορετικά κινδυνεύουμε από πολύ σοβαρά προβλήματα. Στο δεκείμενο εδώ μιλάτε για την απαγόρευση κάποιων συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Γιατί... Λέτε ότι δεν αντιλαμβάνεστε μεν τα επιχειρήματα, αλλά εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω ένα επιχείρημα. Τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι όντως καλή λύση το να απαγορεύουν οι πολιτικοί κάτι, γιατί τελικά ε, κάπου αλλού θα βρεθεί η διέξοδο και η λύση. Δηλαδή μόνο απογορεύσει θα χρειαστούμε να επιβάλλουμε. Θα καταντήσουμε να επιβάλλουμε. Τώρα για τι αρχέ αυτέ. Τι είδου στόχο μπορεί να εξυπηρετούν. Να κάμψουν την αγορά. Να είναι πιο βραδία η λειτουργία της αγοράς. Γιατί να πληρώνουμε τελικά πιο πολλού φόρου. Ε, να βάλουμε νέου φόρου. Και εγώ τι να σα πω, είμαι από χώρα που έχει του ψηλότερου φόρου στην Ευρώπη, στον κόσμο ίσω. Ο φόρο θα πρέπει σιγά σιγά να μειώνεται μάλλον, γιατί δεν θα είναι τα χρήματα διαθέσιμα για πάντα. Και ίσως πέραν της, ε, των φόρων θα πρέπει να δούμε και το περιβάλλον, την αναπτυξιακή βοήθεια, όλα αυτά. Να ευχαριστώ πολύ καλή συζήτηση. Πολύ καλή ερώτηση για τη συζήτηση. Στο έγγραφό μας καθιστούμε σε θέση ότι αντιλαμβανόμεθα τους ε, υπερβολικούς κινδύνους, το γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής ρύθμιση του κινδύνου, διαχείριση του κινδύνου, αλλά η απαγόρευση ορισμένων προϊόντων δεν είναι για μας η λύση. Γιατί τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα από μόνα τους δεν είναι φορείς κάποιας ε, ε, αμαρτίας προπατορικής. Και υπάρχουν ε, κανόνες και για την χειραγώγηση της αγοράς και για την κατάχρηση αγορών Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι υπάρχουν σαν και μπορούμε όπως έγινε και με την Norman Sachs ε, υπάρχουν δηλαδή κανόνες που μπορούμε να τους εφαρμόσουμε για να πατάξουμε την χειραγώγηση των κεφαλαιοχικών αγορών ή για να δώσουμε τις λύσεις εκεί που χρειάζεται. Τα ΣΧΟΠ λοιπόν έχουν κάποια βάση. Το να απαγορεύσουμε ορισμένα προϊόντα δεν μας απαλλάσσει ούτε από τα χρέη, ούτε από τίποτε άλλο. Μάλλον περιορίζουμε περιορίζοντας την νομιμότητα ενός εγγράφου, το καθιστούμε μάλλον ε, πρόσφορο στο hedging, δηλαδή στην ασφάλιση κινδύνου. Και έτσι θα αρχίσουν να βγαίνουν προϊόντα για την ασφάλιση από την απαγόρευση ή της απαγόρευσης. Και νομίζω ότι υπάρχουν ήδη κανόνες, στους οποίους ε, θα έπρεπε απλώς να εφαρμόσουν τα κρατη Εάν δούμε ότι κάποιοι αγορέ λειτουργούν συντονισμένα, πρόκειται για κατάχρηση της πόσες θέση και υπό το ευρωπαϊκό δίκαιο και υπό το βρετανικό τουλάχιστον δίκαιο. Και για τις αγορές των ε, παραγόγων και για πολλές άλλες κατηγορίες δραστηριοτήτων υπάρχουν λύσεις διαφορετικές από το να ε, απαγορεύουμε προϊόντα. Αυτό μόνο την η συνέπεια θα είχε να μειώσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε σχέση με τις εθνείς αγορές. Επίσης, θα θυμάστε το παλαιό μοντέλο του νόμου Τόμπεν στη δεκαετία του 70 και του 80. Και την αδυναμία που προκάλεσε για την άντληση κεφαλαίων σε περιοχή κρίσεων. Στην ενδιάμεση λοιπόν έκθεση προτείνεται φόρος ε, σταθεροποίησης της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας και φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. φόρο αντίστοιχο με τον τόμπενο, όπω όπως φόρο μειώνει παραδείγματι και τέτοια. Το Διεθνέ Νοσηματικό Ταμείο πρόκειται με βάση τη μελέτη του Απριλίου, που δόθηκε πριν από δύο εβδομάδε, να διατυπώσει συμπεράσματα από ό,τι φαίνεται. Οι φόροι πιστεύω θα πρέπει να επιτελούν δύο έργα. Αντικυκλική ρύθμιση, αφενός, φόρος επί των κερδών των τραπεζών, παραδείγματι, σε εποχές παχιών αγελάδων για τις τράπεζες, θα έφερνε πολλά φορολογικά έσοδα. Και σε μια δύσκολη εποχή, την ώρα που το κράτος είναι πιο φτωχό και που οι τράπεζες ενδεχομένως καταραίουν, για να στηριχθούν οι τράπεζες θα μπορεί το κράτος να αντλήσει από αυτήν ακριβώς την ε, φορολογία επαρκή κονδύλια. Μπορεί λοιπόν, εάν εφαρμοστεί σωστά ένα τέτοιο μέτρο ή τέτοια μέτρα, να, φορολογικά δηλαδή, να προσφέρουν ε, αναγεννούμενες πηγές εσόδων και για την ε, αντιμετώπιση της φτώχειας και για τις κλιματικές αλλαγές και για τους στόχους της χιλιετίας. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει οι υπεύθυνοι για, ε, για τη λήψη αποφάσεων φορείς να λάβουν υπόψη αυτή τη λύση της προλογίας, διότι μπορεί να αποτελέσει πηγή μακροπρόθεσμη και για την εξυπηρέτηση μακροπρόθεσμων προγραμμάτων και γενικότερα πραγματικών πολιτικών, πηγή εσόδων η φορολογία. Ο Πρόεδρος. Αν μου επιτρέπετε θα θέλω να φερθώ σε δύο-τρία ζητήματα. Να επανέλθω καταρχάς ε, στο ζήτημα της μόχλευσης. Το συμπέρασμα ότι η ανάγκη για ανάληψη δράση στην Ευρώπη είναι πολύ πιο έντονη από τις ΗΠΑ. Χειρότερα τα πράγματα μάλιστα γιατί δεν υπάρχει τέτοια ομοιογένεια μεταξύ των τραπεζών της πυρωτικής Ευρώπης. Γιατί έχουμε παραδείγμα τις, Ισπανικές και τις Ιταλικές ε, τράπεζας που έχουν ε, επίπεδο μόχλευσης περί το 20% ενώ οι γερμανικές και οι γαλλικές είναι περί το 40%. Και μπορώ να σας πω εγώ για τη Γερμανία που ξέρω ότι υπάρχει και το λεγόμενο εξαρτούμενο χρέος, subordinated debt, και το οποίο επίσης ε, την χάνει χειρισμών αντίστοιχων με αυτών ε, των παραγόγων. Άρα μπορούμε να φτάσουμε σε διψήφια, τριψήφια νούμερα χωρίς να καταλάβουμε πώς μας συνέβη αυτό. Απάντηση. Ναι, έχουμε ένα τρένο το οποίο έχει μπει μέσα και έρχεται να, να συγκρουστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περές. Στο λαιμό σας τα έχετε, τα ναι. ακουστικά. Πριν, ε, γιατί θα ήθελα να ακούσουμε τα στοιχεία που δώσατε, είναι εξωφρενικά. Το ότι μα κοροϊδεύει βέβαια η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών το καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται δηλαδή. Αλλά πώ την εξηγείτε την κατάσταση. Ω εκπρόσωποι και υπεύθυνοι στην Ευρώπη Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, έτσι. 70% χρηματοδοτείται από τι οικονομικέ δραστηριότητε στην Ευρώπη χρηματοδοτείται από τις τράπεζες, αντίθετα από τι ΗΠΑ. Πώ το εξηγείτε αυτό, δηλαδή είναι έξω από τα επίσημα νούμερα, ε, off balance sheet αυτό, αυτή η δραστηριότητα. Ή μήπω στι Αμερικανικέ τράπεζε υπολογίζεται το σύνολο των ε, τραπεζών ή μόνο οι μεγάλε ή μόνο εκείνες που εφαρμόζουν κάποιο συγκεκριμένο σύστημα. Πού έγκυται αυτή η διαφορά, ποιο είναι το μυστήριο, διαφωτίστε μας. Το επόμενο σημείο αναφερθήκατε στο πρόβλημα too big to fail. Πώς να επιληθεί. Ε, είπα το έχει αναλογική αύξηση μόνο, αλλά υπέρ του αναλογικού αύξηση του κεφαλαίου. Συναγάγατε το συμπέρασμα αφού αξιολογήσατε όλα στη δυνατότητε έχουμε συστάσει του ΩΣΑ. Τι λένε. Λένε οι τράπεζε να οργανωθούν ούτω ώστε αν επιχειρήσεις δεν πάνε καλά καταρρεύσουν και πρέπει να εξαλειφθούν η τράπεζα θα πρέπει να είναι οργανωμένη ούτω ώστε οι υπόλοιπε επιχειρήσεις να μπορούν να λειτουργούν. Το εξετάσατε? Συγκρίνατε τα υπέρ και τα κατά των δυνατοτήτων. Πριν καταλήξετε στα συμπεράσματα. Τέλος. Είναι φιλοσοφικό θέμα το τελευταίο. Τι χρειαζόμαστε για να μην την ξαναπατήσουμε. Να αλλάξουμε συμπεριφορά πρέπει. Και η αλλαγή συμπεριφορά είναι το δυσκολότερο πράγμα που μπορεί να περιμένει κανείς από το ανθρώπινο «ον». Ερώτηση τα προβλήματα που εξετάζουμε οι ρύθμιση στη κύματα, κεφαλογικές ε, απαιτήσει, η επιτροπή στιμικού κινδύνου κλπ. Αυτοί οι μηχανισμοί αρκούν, μπορούν να σπάσουν τις κακές συνήθειες ή πρέπει να εφεύρουμε κάτι ακόμα πιο αποτελεσματικό, πιο δραματικό. Απάντηση. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Πώς θα προσαρμοστεί η Ευρώπη στις νέες ρυθμιστικές αλλαγές. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να διεθνεί στους φορείς τυποποίηση στους διεθνείς. Δεν θέλω να αποσυρθεί η Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να επηρεάσει όμως τη συζήτηση περισσότερο από ό,τι τώρα. Διότι οι συνέπειες των προτάσεων Βασιλείας 2 του περασμένου Δεκεμβρίου θα είναι καταστροφικές για πολλά τραπεζικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Ένας από τους λόγους είναι διότι η Συμφωνία Βασιλείας δεν ρύθμισε ποιο πρέπει να είναι το ρυθμιστικό κεφάλαιο, από τι αποτελείται συγκεκριμένα, υποδιαιρέτω σε κατηγορία επίπεδο 1, επίπεδο 2. Και έλεγαν ότι πρέπει να είναι κοινέ μετοχέ, προτιμησιακέ μετοχέ και κάποιο δευτερεύον χρέο κλπ. στο επίπεδο 1. Και οι υποπτικέ αρχέ των 100 μελών έπρεπε αυτά να τερμινεύσουν και τα εφαρμόσουν. Και είχαμε την κατηγορία 2, επίπεδο 2, άλλα ε, αξιόγραφα που ήταν πιο επικίνδυνα και ομόλογα δεν υπήρχε συγκεκριμένο ορισμός τι σήμαιναν όλα αυτά. Και στο τελικό δίκαιο των χωρών ε, δεν υπάρχουν προτιμησιακές ε, ε, μετοχές. Οπότε οι Ελβετοί έχουν διαφορετική προσέγγιση. Στο επίπεδο 1 έχουν απλές μετοχές με κάποιο δευτερεύον χρέος. Σε, σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχει περισσότερα, οι χώρες έχουν περισσότερα μέσα χρέους. Διότι αυτά όμως έχουν λιγότερα δυνατότητα να απορροφήσουν απόλυση όταν αντιμετωπίζει προβλήματα η τράπεζα, ενώ οι κοινέ μετοχές μπορούν να απορροφήσουν καλύτερα ε, το, τις απώλειες. Χάνει, χάνει κανείς ε, τα πάντα χρεοκοπήσει, άμα έχει μετοχές η τράπεζα. Άμα υπάρχουν μέσα χρέους, ε, μπαίνει φερεγκαιότητα μες στο παιχνίδι. Οπότε το κεφάλαιο ε, επίπεδου 1 θέλουν να είναι μετοχέ κεφαλαίου και απορροφά τη ε, απώλεια. Αυτό είναι σημαντικό για την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη παραδοσιακά ε, δεν έχει συμμετάσχει σε Εθνική Συμφωνία για το τι είναι το επίπεδο 1. Έχει διάφορε πρακτικέ που ακολουθεί η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του επίπεδου 1. Άρα οι περισσότερε χώρε τη υπηρετική Ευρώπη έχουν νομοθεσία που προβλέπουν ότι το επίπεδο 1 είναι προτιμησιακές μετοχές, όπως αποκαλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στις ΗΠΑ. Είναι ουσιαστικά μετοχή, αλλά χρέο. Είναι αξίωση. Της, ε, αν η επιχείρηση εκπροποποίηση είναι μια αξίωση, δεν εξαφανίζεται. Ενώ στι ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε πιο απλέ μετοχέ που αποτίζουν το επίπεδο 1. Κατά κάποιο τρόπο είναι πιο εύκολο για τι τράπεζε να μαζέψουν χρήματα εκδίδοντα περισσότερο χρέο που χρηματοδότησε. Χρησιμοποιούν σαν, σαν ρυθμιστικό κεφάλαιο κάποιο αυτό το χρέο. Ε, διότι εκδίδουν περισσότερο χρέος και επενδύουν. Ε, λοιπόν, και είναι πιο δαπανηρό να προσαρμόσει κανεί το ποσοστό μόχλευση. Είναι ένα πρόβλημα εφαρμογή που κατά παρελθόν η Επιτροπή Βασιλεία πάντα υιοθετούσε γενικέ προδιαγραφέ που εφαρμοζόταν ποικίλο τρόπο. Αλλά τώρα λόγω τη κρίσεω λένε τώρα, τώρα ένα από τα προβλήματα είναι ότι οι χώρε δεν έχουν επαρκέ κεφάλαιο. Άρα θα πρέπει να καθορίσουμε τι είναι το κεφάλαιο πάρα πολύ συγκεκριμένα. Οπότε είναι πολύ μεγάλο ζήτημα είναι γιατί ποτέ δεν καθορίστηκε τι είναι το κεφάλαιο, τι θα έπρεπε να είναι συγκεκριμένα προηγουμένω. Άρα αυτό είναι το πρώτο και είναι μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό που θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη θα είναι να προσπαθήσει να, κάνει, να συμμετάσχει στην Επιτροπή τη Βασιλεία και να πει αν θέλουμε να αλλάξουμε τον ορισμό του κεφαλαίου, Α αντικατοπτρίζει λίγο περισσότερο αυτά που κάναμε εμείς στην Ευρώπη. Γιατί θα πρέπει όλα να είναι κοινέ μετοχές των μετόχων. Θα πρέπει να έχουμε και αυτές, αλλά δεν θα πρέπει να είναι απόλυτα έτσι, διότι η ΕΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο το κάνουν διαφορετικά και θα έχουν ε, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τώρα συγκέντρωση και αναλογίε συγκέντρωση. Με ρωτούσατε τι γίνεται αντί να έχουμε περισσότερα τέλη για το κεφάλαιο για τις μεγάλες τράπεζες, μήπως ανταυτού θα πέσουμε να ρυθμίσουμε τις πρακτικές που κάνουμε, να τις ελέγξουμε καλύτερα. Οπότε να μην αφήνουμε την τράπεζα να βασίζεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση υπερβολικά. Να μην έχουμε μια μεγάλη τράπεζα να έχει 80% τη αδειοδότηση στο στεγαστικό τομέα, 60% στις πιστοτικές χρέη πιστοτικών καρτών και αυτό αφορά και τη σύνθεση του στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας. Σε κάποιες χώρες υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη σύνθεση των στοιχείων του ενεργητικού. Μπορεί να έχεις... Δεν μπορείς, παραδείγματος χάρη, να δανείζεις παραπάνω από ένα ποσοστό στην τομέα των κατασκευών. Διότι αν καταρρεύσει ο τομέα των καταδομών, τότε καταραίει και η τράπεζα. Άρα υπάρχουν όρια σχετικά με το πώ εκτίθεσε στου διάφορου κινδύνους των διαφόρων επιχειρήσεων. Και οδηγία και τα κεφαλικές απαιτήσει δίνουν προσανατολισμούς, αλλά έχει συγκεκριμένε απαιτήσει. Είναι καλό που ίσω η Ευρώπη θέλει να έχει περισσότερε συγκεκριμένε απαιτήσει πάνω σε αυτό. Και ίσω οι μεγάλε τράπεζε να είναι πιο ισορροπημένε, το τρόπο στον ΕΒ. Βεβαίω ε, ε, μια τράπεζα χρεοκόπησε 80% των στοιχείων ενεργητικού στη δανειοδότηση στεγαστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Και όταν κατέρευσε το στεγαστικό τομέα, ε, κατέρευσε, έχασε τη χρηματοδότηση τη τράπεζα και κατέρευσε. Χρειάζεται συγκεκριμένοι κανόνε όσον αφορά τη σύνθεση των στοιχείων ενεργητικού τραπεζών, ώστε να μην βασίζονται υπερβολικά σε οδήποτε συγκεκριμένο τρομέα. το κάνετε αυτό, τότε το πρόβλημα του big to fail ίσω να καλυφθεί. Αλλά τώρα οι μεγάλε τράπεζε βεβαίω είναι πάρα πολύ ποικιλόμορφε αφορά τι δομέ του. Άρα η Citigroup, παραδείγματο χάρη, δεν είναι 80% στεγαστικά, οι πιστοτικέ κάρτε 60% επειδή είναι μεγάλες έχουν τα δραστηριότητε, Ίσως να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα τη συνθέσεω των στοιχείων ενεργητικού στι λίγε τράπεζε μεγάλε που είδα. Αλλά υπάρχει στην οικονομική θεωρία και υπάρχει ένα επιχείρημα ισχυρό που λέει ότι επειδή μεγάλε τράπεζε ενδεχομένω δημιουργούν συστημικό κίνδυνο ε, στο big to fail, στο πρόβλημα, θα πρέπει να πληρώσουν γι' αυτό. Και δεν είναι πρόβλημα να πληρώσουν, διότι βγάζουν πάρα πολύ μεγάλα κέρδη και μεγάλε συνεργασίε δημιουργούνται και είναι μεγάλε. Είναι πολύ σημαντικό όμω να μην βασιζόμαστε υπερβολικά σε αυτό. Επίση, δεν ανέφερα ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε και στην πολιτική ανταγωνισμού. Γιατί αυτέ οι τράπεζε γίνονται τόσο μεγάλε, γιατί έχουν τόσο μεγάλο μερίδιο τη αγορά. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ολιγοπόλιο στι τράπεζε. Ε, η αρχή του ανταγωνισμού θα πρέπει να επιβάλλει τον κανόνα, τον το νόμο περί ανταγωνισμού. Ναι, εκτός διάλογος, εκτός μικροφώνου. Και δεν μπορούμε να μαντέψουμε τι λέει η κυρία Πέρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η απάντηση, τέλο πάντων. Δεν ξέρω ποια είναι η λογική που κρύβεται πίσω από αυτό. Υπήρξαν αιτήματα και αυτό είναι επαναλαμβανόμενο θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κανόνε βεβαίω, βεβαίω, όσον αφορά τη συγκεντρώση στην αγορά. Αλλά ουσιαστικά πιστεύω ότι οι νόμοι περί ανταγωνισμού βασικά απαγορεύουν καθορισμό των τιμών και αν υπάρξει μεγάλο μερίδιο της αγοράς, μπορείς να καταχραστείς τη θέση σου στην αγορά. Και αν δείξει ότι η τράπεζα δεν καταχράται τη θέση στην αγορά, συμμορφώνεσαι. Αν δεν καθορίζεις τιμές, αν δεν καταχράσει τη θέση σου στην αγορά, απλώς με το να είσαι μεγάλος, αυτό καθεαυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα. Δεν είμαι ειδικό για το δίκαιο περί ανταγωνισμού, αλλά λέω ότι ενδεχομένω, πιθανώ οι μεγάλε τράπεζε δεν ερευνήθηκαν διότι ο ρυθμιστικός φορέας δεν θεωρεί ότι καταχρώνται τις θέσεις του στην αγορά. Πρόεδρος, Ότμαρ. Λοιπόν, Λοιπόν, δόθηκε η πρόταση, έγινε η πρόταση να κάνουμε έναν ορισμό του κεφαλαίου αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και η Βασιλεία 3 και θα γίνει μια διαβούλευση με τον όσα. Δεν ξέρω, εδώ διαπιστώστε κάποιες διαφορές όσον αφορά τις τράπεζες και το πόσο φύγονται οι τράπεζες. Πού οφείλεται αυτή η διαφορά στο πόσο θίγονται οι τράπεζες. Οφείλεται στην, στον διαφορετικό ορισμό του κεφαλαίου. Έγκυται διαφορά στο ότι αυτός ο ορισμός ανταποκρίνεται περισσότερο στις επενδυτικές τράπεζες και όχι στις, ε, τράπεζες, ε, στις λιανικές τράπεζες. ή έγκυται στο ότι εδώ ε, προσπαθεί κανείς ε, να κάνει μια, να ασκήσει μια πολιτική, μια συγκεκριμένη πολιτική. Δεν ξέρω, ε, η ερώτησή μου έχει ως εξή. τι θα έπρεπε να κάνουμε ούτως ώστε να ξεπεραστεί αυτή η διαφορά. Γιατί εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμία δημοκρατική πλειοψηφία στην Ευρώπη, ούτε στην αγορά, ούτε στο επίπεδο των κοινοβουλίων. Ή για να συμφωνήσουμε με την Βασιλεία Τρία. Η δημοκρατική πλειοψηφία θα κριθεί όταν έχει ολοκληρωθεί η Βασιλεία Τρία. Και αυτό είναι το επόμενο προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ε, τι πιθανότητες ε, βλέπετε εσείς στην Επιτροπή Βασιλείας να επιτευχθεί η υπέρβαση αυτής της διαφοράς μέχρι τον Ιούνιο. Νομίζετε ότι μέσω μιας αξιολόγησης των επιπτώσεων ή μέσω μια αξιολόγηση των επιπτώσεων της ρύθμισης αυτής στην πραγματική οικονομία ως, ε, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια διαφορετική αλλαγή νοοτροπίας πιστεύω θα πρέπει να εντοπίσουμε τα αίτια αυτής της ε, ανισότητας, αυτής της αδικίας, γιατί εάν γνωρίζουμε ποια είναι τα, έννοια, ε, αίτια αυτής της αδικίας, ε, θα απευθυνθούμε στο σωστό παραλήπτη για να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Στην υπάρχουσα βάση δεν θα έχουμε, δεν θα κρατήσουμε δημοκρατική πλειοψηφία για τα αποτελέσματα της Επιτροπής της Βασιλείας παρόλο που πραγματικά θέλουμε να επενδύσουμε όλα στην ενίσχυση των κεφαλαικών απαιτήσεων για να αποκριθούμε σωστά στην κρίση. Εάν ε, δεν ε, ε, μπορέσουμε να πετύχουμε μια συμφωνία, θα υπάρξει μια απόλυτη εμπιστοσύνη όσον αφορά τις πολιτικές αντιδράσεις, την πολιτική απάντηση στην παρούσα κρίση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση θα πρέπει να δούμε τα επίπεδα κεφαλαιοκών απαιτήσεων με τα οποία πρέπει να υπάρχει συμβατότητα. Νομίζω ότι η λύση για την ευρωπαϊκή κοινότητα είναι να ξεκινήσει το διάλογο με την Επιτροπή της Βασιλείας, η οποία βασίζεται σε μια συνένεση και δεν θα οριστικοποιήσουν καμία συμφωνία εφόσον υπάρξει, παρά μόνο εφόσον υπάρξει μια συνένεση. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα επενδύσουν πολύ περισσότερα κεφάλαια στις τράπεζές τους για να μπορέσουν να είναι συμβατές με τις προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας. Ωστόσο αυτές οι προδιαγραφές είναι αντικείμενο συζήτηση, αντιπαράθεση. Ίσως το φθινόπωρο θα αλλάξουν ε, γιατί η Γερμανία συμμετέχει στην Επιτροπή Βασιλείας και λοιπά και ενδεχομένως και άλλες χώρες μπορεί να επηρεάσουν τη συζήτηση. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχει τέτοιες επιπτώσεις. Αλλά έστω και αν υπάρξει επιτευχθεί ένα συμβασμό και έχετε δίκιο, αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια απλή πρόταση που λέει εάν έχουμε υψηλά επίπεδα κεφαλαίου ε, και από την άλλη υπάρχουν ε, απλές, έχουμε απλές μετοχές. Τι θα πρέπει να γίνει. Ε, δεν ξέρω, θα πρέπει το κεφάλαιο να συντίθεται από μετοχές. Ε, δεν ξέρω, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα μέτρα, η πιστοτική κίνδυνη η κρίση δεν ε, προκλήθηκε από κεφαλαϊκή ανεπάρκεια, αλλά από προβλήματα ρευστότητας ε, στο σύστημα. Αυτό έκανε το σύστημα να καταρρεύσει. Λέγοντας λοιπόν ότι ας έχουμε υψηλότερα επίπεδα κεφαλαίου και ως μερίδια μετοχών, το κεφάλαιο, αυτό δεν μπορεί να απειλήσει το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα είναι πρόβλημα ρευστότητας μπορούμε να πούμε ότι και η Βασιλεία 2 οδηγεί τις τράπεζες σε χαμηλά επίπεδα κεφαλαίου. Και αυτή τη στιγμή ξεσπάσει η κρίση, θέλουμε οι τράπεζες να είναι παρακώς κεφαλοποιημένες για να μπορούν να απορροφήσουν τα σοκ λόγω της ύφεση. Αλλά πρόκειται για ένα σχεδιασμό, δεν μπορούμε να να αυξήσουμε τα επίπεδα του κεφαλαίου και να γίνει όλο το κεφάλαιο μερίδια μετοχών. Θα πρέπει να έχουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση, να λέω ότι έχουμε υψηλότερα κεφάλαια, να έχουμε ε, μερίδια μετοχών, αλλά να προσεγγίσουμε και τα προβλήματα ρευστότητας στην ε, αγορά τιτλοποιημένων, ε, στην αγορά των τίτλων. Ε, και να δούμε τι γίνεται και με τα ομόλογα. Εάν θα πρέπει να πάνε στα, στους οργανισμούς συμψηφισμού για τι είναι δυνάμει σε θέση να απορροφήσουν τους κινδύνους και τα σοκ. Οι οργανισμοί συμψηφισμού βεβαίως συνδέονται με προβλήματα ρευστότητας. Και αυτό είναι το τμήμα της αγοράς που μας οδήγησε στην κρίση το 2007. Δεν ήταν η μικρή ε, κεφαλοποίηση των ε, τραπεζών. Και οι τράπεζες πρέπει να έχουν, ένα, έχουν ψηλό κεφάλαιο. Η Επιτροπή Βασιλείας ασχολείται τώρα με το θέμα αυτό. Αλλά αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση εν σχέση με το πώ ρυθμίζουμε το συστημικό κίνδυνο το ζητούμενο, ε, ε, όλα αυτά δεν είναι γύρω από τις αναλογίες μόχλευσης και το τραπεζικό κεφάλαιο, αλλά τη διάρθρωση της ρευστότητας στις χρηματαγορές και στις ε, αγορές κινητών αξιών. Εκεί επέτυχε η αγγλοαμερικανική προσέγγιση και κατέρευσε, γιατί δεν είχαν μια τέτοια διαφορεμένη αγορά στη Γερμανία ε, που να αγοράζει τυλοποιημένα προϊόντα από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Η τυλοποίηση έγινε στις ΗΠΑ ε, και στο, στη Μεγάλη Βρετανία και αυτό είναι το συστημικό κινδύνου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το συστημικό κίνδυνο από διάφορες προοπτικές γωνίες και νομίζω ότι η Επιτροπή Βασιλείας το εξετάζει από μία γωνία που αφορά το τραπεζικό σύστημα. Ε, γι' αυτό θα σύστηνα στην Ευρώπη μία πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση. υπήρξε μια ερώτηση προηγουμένως, κυρία μου, σε σχέση με το πώς θα είναι η μελλοντική χρηματοδότηση. Θα πρέπει να υπάρξουν αυτές οι κεφαλαϊκές απαιτήσει. Ποια είναι η λύση. Ορισμένες χώρες νομίζω θα πρέπει να εξετάσουν ιδιαίτερα εκείνες που δεν έχουν διαρθωμένες αγορές, χρηματαγορές όπου όταν βασίστε περισσότερο σε τραπεζική χρηματοδότηση και έχετε εθνικές ε, τράπεζες που επιδοτούνται από τους φορολογούμενους και κάνουν ε, μακροπρόθεσμα δάνεια. Στην ε, Ελβετία οι τράπεζες επιδοτούνται από τους φορολογούμενους. Μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στη Ζηρίχη και εξαιρούνται από το, νόμο, από το Ευρωπαϊκό Νόμο περί ανταγωνισμού. Εάν θέλετε να αναπτύξετε τις εθνικές σας τράπεζες, θα πρέπει να βρείτε ένα τρόπο αυτό να είναι συμβατό με τον Ευρωπαϊκό Νόμο περί ανταγωνισμού. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει αναπτύσσοντας τις οικονομίες της αγοράς. Στην Ελβετία έχετε μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες, UBS της Ελβετίας, όπου έχετε ένα συνδυασμό μεσαίων τραπεζών που οι ιδιοκτήτες είναι τα καντόνια και έχετε και ιδιωτικέ τράπεζε, μικρέ, ιδιωτικέ τράπεζε και μεγάλε ε, δημόσιες, ε, εθνικές τράπεζες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν άλλε ερωτήσει. Ναι, ναι, αντιδράσω αυτή τη τελευταία πρόταση, βέβαια μου αρέσει και είναι και σύμφωνα με πρωτοβουλίες που έχουν λάβει και το Ίδρυμα Μαργκριτ και άλλοι. Είναι θέματα ανοιχτά και με το Ηνωμένο Βασίλειο που ο Νίκ Κλέκ έκανε κάποιες προτάσεις που θυμίζουν λίγο τέτοιες ανησυχίες σαν αυτές που, είπατε, που εκφράσατε κι εσείς αλλά το θέμα δεν είναι μόνο οι τράπεζε κάνουν τη δουλειά του, όπως είπατε. Αλλά πώς θα εξασφαλίσουμε ότι όλες οι τράπεζες θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουν ναι, δεν είναι μόνο να κερδοσκοπούν και να δημιουργούν ε, φούσκε. Πώς λοιπόν όταν χρησιμοποιούν τα χρήματά τους τα χρησιμοποιούν για να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία και όχι για να κατασκευάσουν νέε σαπουνόφουσκε. Την πρόταση βεβαίω και τη δέχομαι, είναι εύκολο. Να σας πω, η πρόταση Βόκερ, παραδείγματι, που έχει τώρα ενστερνιστεί ο Ομπάμα στις ΗΠΑ. Τράπεζες οι οποίες έχουν εγγυηθεί από θέματα δεν μπορούν να μπουν στις, ε, στην χρηματοπιστωτική αγορά για δικό τους λογαριασμό, μόνο για λογαριασμό των πελατών τους. Και άρα, εάν δεν θέλει να πάρει αυτήν την εγγύηση αποθεματικού από το κράτο, κάνει ό,τι θέλει η τράπεζα. Αλλά με την ε, πρόταση Βόκερ, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα πιστεύω, διότι δεν βλέπω να μπορεί να αντιμετωπίσει τον συστημικό κίνδυνο μεν, πλην όμως θεωρώ ότι ορισμένες τράπεζες ίσως να εξαρτηθούν λιγότερο ε, ίσως να εξαρτηθούν λιγότερο από τις επενδύσεις τους στον κίνδυνο και ίσως να γυρίσουν στις παραδοσιακές τραπεζικές λειτουργίες συμβουλευτικό ρόλο σε σχέση με κάποιου πελάτε κτλ. Δηλαδή περιορίσουν το πεδίο δράσεών του και ίσω τελικά να είναι πιο ασφαλεί και πιο σταθερέ. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε τι μεγάλε επενδυτικέ τράπεζε που τώρα λαμβάνουν κίνδυνο. Θα υπάρχουν πάντα, αλλά τουλάχιστον θα έχουν τη σχετική ασφάλιση και δεν θα επιδοτούνται από το φορολογούμενο. Εγώ δεν λέω βέβαια ότι θα πρέπει να ακολουθήσει το σύστημα ε, Βόκερ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό καθεαυτό απλώς είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξουμε και θα πρέπει λίγο πολύ οι τράπεζες να περιορίσουν το επιχειρησιακό τους πρότυπο, να έχουν πιο περιορισμένο ε, πεδίο δράσης, πελατολόγιο, και δραστηριοτήτων ε, πεδίο και μετά θα υπάρχουν μεγάλες, η Deutsche Bank του κόσμου, οι οποίες θα κάνουν τις επενδύσεις τις μεγαλεπίβολες, αλλά από την άλλη θα έχουν πιο αυστηρό κίνδυνο, πιο αυστηρό έλεγχο και δεν θα ε, έχουν και την εγγύηση του κράτους για τους κινδύνους που αναλαμβάνουν. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενημερωτικά τα όσα μας είπατε. Συνεχίσαμε τη συζήτηση νομίζω Σας ευχαριστώ όλους αγαπητοί συνάδελφοι και τους διερμηνείς που αντέξανε. Ήταν φρικτό αυτό το απόγευμα. Το ξέρω. Κύριε το πέρα της συνεδριάσεως. 6 Μαΐου η προσεχής. Για να συνεχίσουμε τη συζήτηση στο τελευταίο έγγραφο εργασία